Καλημέρα. Καλημέρα σας. Είναι 9 και τέταρτο. Κομίση Παρλαμέντου Ευρωπαϊκού και Και ξεκινάμε τη δεύτερη μέρα της συνεδρίασης της Επιτροπής ΙΜΚΟ και των Εθνικών Κοινοβουλίων την κοινή συνεδρίαση για την ενιαία στρατηγική της εσωτερικής αγοράς. Και θα συζητήσουμε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις αυτού του θέματος. Σήμερα θα συζητήσουμε τη διακυβέρνηση, την ηγεσία, την ε, συνεργασία, εταιρική συμμετοχή και την ενδυνάμωση. Θέλω να καλωσορίσω όλους τους εκπροσώπους των Εθνικών ε, Κοινοβουλίων, των, τους Ευρωβουλευτές, τους, ε, τα μέλη της Επιτροπής ΙΜΚΟ, της οποίας πρόεδρος είναι ο κύριος Χάρμπορ και σας υπενθυμίζω τη διαδικασία της συνεδρίασης. Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι που θέλουν να λάβουν το λόγο πρέπει να συμπληρώσουν αυτό το φύλλο ε, με το όνομά τους, αυτό το μπλε φύλλο, ε, για να ξέρουμε τι θέλουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Και έχουν, έχουμε δώσει τις ε, κάρτες επί τη βάση των αιτήσεων που λάβαμε και έχουμε και έναν κατάλογο ομιλητών. Ε, βάσει των ε, κατευθυντηρίων γραμμών με τις οποίες κάνουμε πάντοτε αυτές τις συνεδριάσεις. Δηλαδή θα μιλάνε δύο εθνικοί βουλευτές και ένας ευρωβουλευτής. Η διάρκεια της παρέμβασης είναι τρία λεπτά για τον κάθε ομιλητή και θα σε ένα μέρος της... Α, θα πρέπει να ρίχνετε ένα βλέφαρο στην οθόνη για να δείτε πόσο χρόνο πέρασε από την ομιλία σας. Παρακολουθείτε λοιπόν ο χρόνος ηλεκτρονικά. Επίσης υπάρχει διαδικασία της μπλε κάρτες, της μπλε κάρτας, όπου την οποία μπορείτε να σηκώσετε διανατάσεως της χειρός για να ρωτήσετε μία ερώτηση που έχει σχέση με την προηγούμενη παρέμβαση, με τον προλαλήσαντα. Και ο ο μιλητής, εις τον οποίο απευθύνθηκε η ερώτησή σας, έχει 30 δευτερόλεπτα να απαντήσει. Szanowni Państwo, Κυρίες και κύριοι, έχουμε προβλέψει τη συζήτηση μέχρι τις 10 και θα ήθελα τώρα να καλέσω την κυρία Καλονιέτε, η οποία είναι η εισηγήτριά μας και μέλος της Επιτροπής ΙΜΚΟ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κυρία Σάντρα Καλιέντε για να κάνει μια σύντομη εισαγωγή στην διακυβέρνηση, εταιρική συμμετοχή και ενδυνάμωση ε, της εστερικής αγοράς. Όχι, Α, δεν έχει. μόνο. Ευχαριστώ. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη που βρίσκομαι σήμερα εδώ στην κοινή συνεδρίαση Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι είναι ο μόνος τρόπος να βρούμε μια καλύτερη λύση, μια καλύτερη λύση για, για τη λειτουργία της κοινής αγοράς, για τη λειτουργία της κοινής αγοράς. Ε, σήμερα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και να βρούμε νέες θέσεις εργασίας επιλύοντας ε, μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Έχουμε τεράστια εμπόδια μπροστά μας και πολλές φορές αποτυγχάνουμε. Αποτυγχάνουμε ε, και μακροπρόθεσμα. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις πιο μακροπρόθεσμες και αποτυγχάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε μαζί για να βοηθήσουμε την εσωτερική αγορά. Όσον αφορά τη διακυβέρνηση και την εταιρική συμμετοχή στην κοινή αγορά, στην ενιαία αγορά, ε, πιστεύω ότι το βασικό μας έργο είναι να εξασφαλίσουμε το υψηλότερο επίπεδο πολιτικής διακυβέρνησης. Αυτή είναι μια πολιτική βούληση την οποία πρέπει να ασπαστούμε για να δυναμώσουμε την ενιαία αγορά και ο πρόεδρος ε, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Κομισιόν πρέπει να συντονίσουν τις ενέργειές τους ε, προς αυτό το στόχο. Διαφορετικά, πολλοί από τους στόχους μας για την ε, εξασφάλιση μιας νέας οικονομικής ανάπτυξης και για την ενίσχυση της αγοράς εργασίας θα μείνουν μόνο στα χαρτιά και δεν θα μεταφραστούν σε έργα. και θα πρέπει η Ευρώπη να ξαναγίνει α, να μην ε, αποτύχει σε διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό χρειάζονται άμεσες δράσεις μπορούμε να μιλήσουμε για εθνικές ε, δράσεις για τη βελτίωση των εσωτερικών αγορών. Αλλά χωρίς μια συντονισμένη δράση δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε πλήρως την ενιαία αγορά. Έχουμε καλέσει, έχουμε ζητήσει με εξαίσθηση και ψηφίσματα και μέσω του Προέδρου μας και των μελών να, βρεθούν λύσεις το ταχύτερο δυνατόν. Υπάρχουν τομείς όπου αναμένουμε την Κομισιόν να αναλάβει δράσεις μετά το καλοκαίρι, την καλοκαιρινή διακοπή. Καταρχάς την ενιαία ψηφιακή αγορά, εκεί αναμένουμε πρόοδο, ε, ε, την, διανοητική ή πνευματική ιδιοκτησία, ε, τον τομέα της κινητικότητας και την ε, κινητικότητα των αγορών υπηρεσιών, ε, την, ε, επίσης τις αγορές προμηθειών. Σε αυτούς τους τομείς περιμένουμε δράσεις. Τώρα, για την διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή των νομικών, των νομοθετικών μέτρων. Πρέπει να εξασφαλιστεί η μεταφορά και σωστή εφαρμογή των μέτρων αυτών και η Κομισιόν πρέπει να είναι ο θεματοφύλακας και να επιβλέπει αυτή την εφαρμογή. Δεύτερον, πρέπει να μειώσουμε τις τάσεις του προστατευτισμού, διότι ο προστατευτισμός μόνο το μόνο που κάνει είναι να διασπά, να διασπά και να βλάπτει την ανταγωνιστικότητα της ενιαίας αγοράς. Τρίτον, πρέπει να μειώσουμε το κόστος διαφορετικών, διαφόρων ε, τομέων. Ε, Παραδείγματο χάρη τις εξοδικαστικές ε, λύσεις ε, επιλύσεις ε, διαφορών. Να μειώσουμε το κόστος αυτών, το, αυτού του τομέα. Και ε, τέλος πρέπει να βοηθήσουμε, να ενισχύσουμε την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Για, γι' αυτό είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί το πρόγραμμα δράσης σύμφωνα με τις αρχές της Συνθήκης Λισαβόνας. Θέλω να καλέσω τους να ζητήσω από τους εθνικούς βουλευτές να αναλάβουν ε, περισσότερη δράση, να είναι πιο ε, επίμονοι ε, στην ενεργοποίηση αυτών των, των μέσων για να αλλάξει αυτή η κατάσταση που ενημερωπίζουμε σήμερα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί και μάλιστα δραστήρια διότι όλοι οι πολίτες μας σήμερα αναμένουν μία ενεργό συμμετοχή, ε, δική μας δηλαδή συμμετοχή, στην εξέβρεση λύσεων. Εάν καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε και να βελτιώσουμε η λειτουργία της ενιαίας αγοράς, θα προσφέρουμε μια νέα βάση ανάπτυξης. Και πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Από αυτή την πλευρά, ε, ο ρόλο τη αμοιβαία επικοινωνία μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικό, αλλά και από πλευρά Επιτροπή είναι ε, σημαντικό να κάνουμε αυτή την αναφορά. Υπάρχει σημαντική έλλειψη γνώσεων ε, και ενημέρωση από πλευρά του κοινού και γι' αυτό θα πρέπει και τα Εθνικά Κοινοβούλια να ενημερώσουν την κοινή γνώμη. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο Έχω λάβει τον κατάλογο ομιλητών. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να προσκαλέσω και τους ε, καλεσμένους μας εκτός Βρυξελών ε, να πάρουν το λόγο, γιατί προς το παρόν είναι μόνο βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν ζητήσει το λόγο. Κύριε Γιωχάνσεν. Σουηδία. Α, η κυρία Γκέπχαρτ. Μέλος του Ευρωκοινοβουλίου. Εντάξει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ελπίζω να ακούσουμε τις απόψεις αυτού του σημαντικού θέματος από τους συναδέλφους. Θέλουμε, ε, ή μάλλον ε, κάνουμε πολιτική, είμαστε πολιτικοί εκπρόσωποι των πολιτών και γι' αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο να ενεργούμε στα δικά μας, ε, στους δικούς μας θεσμούς, στα θεσμικά όργανα, αλλά να συνεργαζόμαστε κιόλας. Γι' αυτό, στο θέμα της διακυβέρνησης, το πιο σημαντικό είναι η διαφάνεια. Η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και η διαφάνεια στις αποφάσεις που λαμβάνονται. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσδίδει ιδιαίτερη αξία στο θέμα της διαφάνειας. Και γι' αυτό όταν προετοιμάζουμε νομοθετικά μέτρα είναι πολύ σημαντικό να ακούμε την κοινωνία των πολιτών, να ε, ακούμε και να παρακολουθούμε τις απόψεις, τις ιδέες τους και τις αντιδράσεις τους για να ξέρουμε ανα πάσα στιγμή τι θέματα τους καίνε, τι θέματα τους ενδιαφέρουν, τι θέματα σε ποια, ποιες είναι οι προσδοκίες τους, οι ελπίδες τους και για να μπορούμε να ενσωματώσουμε ε, τις αντιδράσεις και τις απόψεις της κοινωνίας των πολιτών. Ε, με κοινωνία των πολιτών ενώ ε, συνδικαλιστικές οργανώσεις, οργανώσεις καταναλωτών, οι οποίες έχουν πολλά σημαντικά πράγματα να μας πούνε και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να συνεργαζόμαστε και να τους ακούμε και ο κοινωνικός διάλογος είναι πολύ σημαντικός. Όταν μιλάμε για διαφάνεια, εννοούμε και έλεγχο, έλεγχο, εποπτεία, ε, έλεγχο του νομοθετικού έργου, εποπτεία και έλεγχο της ε, μεταφοράς και εφαρμογής του στα εθνικά δίκαια και σε αυτό το ρόλο τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να δραστηριοποιηθούν. Είναι πολύ σημαντική η, ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων σε αυτή την ε, μεταφορά και εφαρμογή, γιατί θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη σωστή εφαρμογή του νομοθετικού μας έργου. Ε, από ό,τι ξέρουμε και έχουμε πληροφορηθεί σε πολλά κράτη-μέλη ή έχει γίνει ελλειπής εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή εσφαλμένη. Γι' αυτό υποστηρίζουμε πάντοτε την ε, Κομισιόν όταν ζητάει αυτή την συγκριτική, το συγκριτικό πίνακα ε, εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη για να μπορέσει να ελέγξει τι και πώς έχει εφαρμοστεί. Υπάρχουν μερικά κράτη-μέλη τα οποία εναντιώνονται σε αυτή την ταμπέλα, ε, σε αυτόν τον πίνακα συγγνώμη, συσχετισμού ε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εναντιώνονται, γιατί έχουν τέτοιες αντι, αντιρρήσεις. Αυτός ο πίνακα συσχετισμού της νομοθεσίας και σύγκριση διευκολύνει την εποπτεία του νομοθετικού έργου και την εφαρμογή, τη σωστή εφαρμογή του στα εθνικά δίκαια. Και τέλος, για να μην, γιατί έχω ήδη ξεπεράσει το χρόνο ε, ομιλία μου, Χρειαζόμαστε ε, μια καλή εσωτερική αγορά, μια αγορά που λειτουργεί σωστά χωρίς προστατευτικά μέτρα, χωρίς προστατευτισμό. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίσουμε το δικαίωμα της εργασίας και την προστασία των καταναλωτών. Αυτές οι δύο πτυχές να λειτουργούν σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Έτσι μόνο μπορούμε να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία των πολιτών προς εμάς. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα παρατηρήσή σας. Βεσλούντα από τη Σουηδία. Ευχαριστώ. Πράγματι, εδώ βρισκόμαστε όλοι γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η εσωτερική αγορά. Σε μεγάλο βαθμό μιλάμε για τον τρόπο ε, με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα αυτή η εσωτερική αγορά. Στην Κροκοβία ε, είδαμε πώς ε, έχουν υπάρξει εμπόδια που ουσιαστικά έρουν τη φύση της εσωτερικής αγοράς δεν μπορούμε να αποδεχτούμε μια κατάσταση όπου έχουμε την Ευρω... το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή που ουσιαστικά μα λένε τι να κάνουμε στα εθνικά κοινοβούλια. Ειλικρινά αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα και ε, θα μας δυσκολεύσει πολύ κατά την οικοδόμηση της ε, ενιαίας αγοράς. Από την άλλη, χρειαζόμαστε έναν συνεχιζόμενο διάλογο και χρειαζόμαστε ξεκάθαρη ηγεσία από, από αυτή την πλευρά. Εγώ είμαι σοσιαλδημοκράτης και πρέπει να πω ότι δεν συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω να μας καθοδηγούν και να μας λένε δηλαδή τι να κάνουμε. Πρέπει να υπάρχει αμφίδρομος διάλογος. Η αποφυγή του προστατευτισμού. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς ε, ο προστατευτισμός αυξάνεται στην Ευρώπη και θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συνδιάσκεψη μόνο και μόνο γι' αυτό γιατί υπάρχουν πολλά παραδείγματα που ανακύπτουν ε, παντού. Δεύτερον, μιλήσατε για την μείωση των δαπανών. Η απλοποίηση των κανόνων ε, για τις μικρές και μισές επιχειρήσεις, καλό μέτρο, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε κάνει και πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά την ε, μείωση των κανόνων και ρυθμίσεων, ούτε έχουμε κατεβάσει το κόστος στην αγορά. Ε, πολλά λέγονται, αλλά στην πράξη δυστυχώς ε, λίγα συμβαίνουν. Έτσι δεν ε, έχουμε πετύχει και πολλά σε αυτό το τομέα. Τώρα, στα διπλώματα τεχνίας, Κατά τη γνώμη μου αυτή ήταν μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για πολλές ε, προεδρίες ε, τα τελευταία 15 χρόνια. Ήταν στην κορυφή του θεματολογίου μας για τόσα πολλά χρόνια και τώρα τελικά καταφέραμε να βρούμε μια λύση. Αυτό δείχνει ότι κάποιες φορές ε, πρέπει να βρούμε μαζί λύσεις. Είναι δύσκολο γιατί είναι, έχουμε το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κανεί δεν μπορεί να πει εγώ έχω 100% δίκιο και σε έχει άδικο. Από την άλλη αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα διάλογο και πάλι ε, στον οποίο θα συμμετέχουν τα διάφορα κοινοβούλια και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι, πράγματι για τα διπλώματα βιστεχνίας Ίσως κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας ε, να σημειώσουμε κάποια πρόοδος προς αυτό. Τώρα, να δώσω το λόγο στον Τζαν Κάρλο Αμελίνη. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Αυτό της όλης διαχείρισης και της εταιρικής σχέσης ε, έχει ιδιαίτερη σημασία για την εσωτερική αγορά και την επικράτησή της, το θρίαμβό της. Ε, θα τονίσω μερικά στοιχεία που μου φαίνονται σημαντικά. Τώρα ακριβώς που έχουμε αυτή την οικονομική κρίση, η οποία θέτει σε δυσκολία την ενιαία αγορά, γιατί έχουμε οθήσει προστατευτικές και το είπαμε ήδη ότι αυτές είναι πολύ έντονες ε, πιεστικές. Ε, και τώρα η κύρια λειτουργία λοιπόν όλων αυτών που πρέπει να γίνουν ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλέπουμε ότι υπάρχει μια αντίθεση. Θα πρέπει όμως ε, διάφοροι να συμμετάσχουν να διευρυνθεί αυτός ο διάλογος ο ευρωπαϊκός και κυρίως ο κοινωνικός διάλογος. Ε, δεν υπάρχουν όμως αρκετοί από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτό το διάλογο ουσιαστικά αποκλείονται από αυτόν τον κοινωνικό διάλογο που συμμετέχουν μόνο οι μεγάλες βιομηχανίες και οι μεγάλες συνδικανιστικές ενώσεις και 20 εκατομμύρια μικρομεσαίες και μικρές μικρές επιχειρήσεις δεν συμμετέχουν ουσιαστικά είναι μόνο θεατές όπως το είδαμε και χθες και στον κόσμο αυτό των μικροεπιχειρηματιών. Εκεί υπάρχουν ελπίδες ε, ώστε να μπορέσουν αυτοί να συμμετάσχουν, να σημειωθεί μια σύγκληση και μάλιστα με μια ιδιαίτερη οικονομική κίνηση, όθηση στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς. Οι κύριοι στόχοι που τονίστηκαν νομίζω ότι είναι ορθοί. Θα πρέπει όλα αυτά να τα προσδιορίσουμε βάσει παρεμβάσεων ενισχυμένων πολιτικών και να έχουμε τη δύναμη να μπορέσουν όλα αυτά να γίνουν δεκτά από τα διάφορα κράτη-μέλη και με ρυθμίσεις ευρωπαϊκής φύσεως περισσότερες και όσον αφορά τον ανταγωνισμό όπως επίσης ε, πώς θα αντιδράσουμε στην προστατευτισμό στην αγορά και με ένα πρόγραμμα δράσης που θα συνδυάσει τις διάφορες εθνικές νομοθεσίες. Σας λέω μόνο ορισμένα στοιχεία από όλα αυτά που θα πρέπει και πάλι να εκτιμηθούν και μάλιστα να εκτιμώνται διαρκώς, όπως ε, οι ρυθμίσεις ε, οι φορολογικές που έχουν τρομερή σημασία για τον εσωτερικό ανταγωνισμό όπως επίσης και για την όλη ροή αυτή και για τον ίδιο τον ανταγωνισμό όπως είπαμε και οι ρυθμίσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζόμενους όλα αυτά είναι απαραίτητα για να μην έχουμε στρεβλώσεις της αγοράς ενάντια στον ενταγωνισμό και στους εργαζόμενους. Και ένα τελευταίο σημείο σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές. Θα ήθελα να παροτρύνω για περισσότερη βοήθεια στις γραμμές αυτής δράσης με μια οδηγία ευρωπαϊκή, το Small Business Act, αυτό που έχει να κάνει με τις μικρές επιχειρήσεις που πρέπει να παίζουν κύριο ρόλο απέναντι και στα ίδια τα κράτη στο δημόσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την παρέμβαση από την Ιταλία. Είναι αλήθεια ότι η εκπροσώπηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντική. Και Πιστεύω ότι μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις εκπροσωπούνται συνήθως ε, ε, ικανοποιητικά, ενώ υποεκπροσωπούνται ή εκπροσωπούνται λοιπόν, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό συμβαίνει στις περισσότερες χώρες, στα περισσότερα κράτη-μέλη και όπως είπατε αυτές οι μικρομεσαίες είναι σημαντικές για την οικονομία μας διότι είναι ευέλικτες και γι' αυτό είναι σημαντικό να τις ενισχύσουμε και να ακούγεται τη φωνή τους. Και τώρα ο κύριος Μπουσόη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκουμε εδώ για την κοινή αυτή συζήτηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια για τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς. Στην Κρακοβία την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο φόρουμ της ενιαίας αγοράς. Ε, θέλουμε όλοι να λειτουργεί ομαλά η ενιαία αγορά. Εγώ θέλω να τονίσω ένα σημαντικό θέμα, τη μεταφορά της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς. 0,9 ήταν το έλλειμμα της μεταφοράς της νομοθεσίας το 2010, αλλά το 2011 ανέβηκε το ποσοστό αυτό σε 2,1% και χωρίς μία έντονη δέσμευση για τη σωστή υλοποίηση και μεταφορά του νομοθετικού δικτύου του νομοθετικού πλαισίου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να υποφεληθούν ε, της ενιαίας αγοράς. Πρέπει λοιπόν ε, να αναλάβουμε τις νέες εντολές, τις νέες νομοθετικές εντολές που μας δίδεται από, την, από τους πολίτες. Πρέπει να δημιουργήσουμε μία σταθερή και ισχυρή συνεργασία μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την νομοθετική διαδικασία και αυτό συμπεριλαμβάνει και την πτυχή της μεταφοράς και εφαρμογής. Ήθελα να τα πω αυτά ε, με την ευκαιρία αυτής της κοινή συνεδρίασης ε, με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ζητώ λοιπόν από τα Εθνικά Κοινοβούλια να αναλάβουν με, εξαιρετική σοβαρότητα ε, και να εξετάσουν το θέμα της μεταφοράς της κοινοτικής νομοθεσίας, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα εθνικά δίκαια. Πολλέ φορέ ομολογώ ότι η μεταφορά αυτή είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Όμως, αν ενισχύσουμε τη συνεργασία μας και την επικοινωνία μας, μεταξύ των θεσμικών οργάνων μας μπορούμε να βελτιώσουμε το αποτέλεσμα της μεταφοράς αυτής. Ένα άλλο σύντομο θέμα είναι αυτοί οι πίνακες συσχετισμών, οι συγκριτικοί πίνακες αυτοί οι πίνακες θα προσδώσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία μεταφοράς και θα μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και οι πολίτες. Επίσης θα υπάρχουν εθνικοί δικαστές οι οποίοι θα κρίνουν την εφαρμογή και θα υποπτεύουν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι συγκριτικοί πίνακες, οι πίνακες συσχετισμών θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν, να εφαρμοστούν ε, γιατί με τον τρόπο αυτόν θα μπορέσουν τα εθνικά κοινοβούλια να πιέσουν τις κυβερνήσεις τους να επιταχύνουν ή να βελτιώσουν την εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. νομοθεσίας. Ξέρω ότι μερικά κράτη-μέλη δεν το επισημούν, δεν είναι διόλου ευτυχή με αυτή την ε, ιδέα. Και τέλο, εφόσον εμεί εκπροσωπούμε τους ε, πολίτε μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη επικοινωνία μεταξύ εταιριών του επιχειρησιακού κόσμου δηλαδή και των πολιτών για τα ωφέλη της ε, ενιαίας αγοράς. Ε, και επίσης θα πρέπει να υπάρξει κάποια ταχεία αντίδραση όταν κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη σχέση συνεργασίας. Ε, πρέπει να υπάρχει μια ταχεία ενημέρωση, ταχεία αντίδραση, διόρθωσης ε, σφαλμάτων και στρεβλώσεων. Γι' αυτό πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων σε αυτή τη διαδικασία της ενιαίας αγοράς, ολοκλήρωσης και βελτίωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την επικοδομητική σας ε, παρέμβαση και Ασφαλώς χρειάζεται μια συνεχής και μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού, ιδίως ε, όσον αφορά την νομοθεσία της ενιαίας αγοράς. Αυτή η συνεργασία είναι λίγα σημαντική και πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν. Έχουμε να κάνουμε πολλά. Ας μην ξεχνάμε και το lobbying που μπορεί να γίνει, δηλαδή η άσκηση πίεσης από ενδιαφερόμενες ομάδες τα εθνικά κοινοβούλια για την πρόωθηση της ενιαίας αγοράς. Τα ωφέλη της ενιαίας αγοράς ε, τα συζητήσαμε ε, εν μέρη και χτες και υπόθηκε ότι πρέπει να βελτιωθεί η επικοινωνία με τους πολίτες μας. Πρέπει να ενημερώνουμε καλύτερα τους πολίτες μας για τα ωφέλη της ενιαίας αγοράς. Τι μπορούν να κερδίσουν από αυτήν, ε, ποια νομοθετικά μέτρα προβλέπει, Γενικώ τα ωφέλη δηλαδή πρέπει να μεταδίδονται στους πολίτες ε, με έναν τρόπο καλύτερης επικοινωνίας. Ο πρόεδρος της ΙΜΚΟ, κύριος Χάρμπορ, έχει κάνει πολλά. Η επιτροπή του ΙΜΚΟ είναι λίγο ορατή και προβάλλεται συχνά στο διαδίκτυο, ε, σε, ε, σε εκστρατείες προβολής των, της ενιαίας αγοράς κλπ. Είναι μη στρατηγική πάρα πολύ καλή που ε, μπορεί να την ε, μιμηθούμε, να την ακολουθήσουμε και εμείς στην Πολωνία. Παραδειγματική λοιπόν ε, στρατηγική για μας. Και τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον εκπρόσωπο της Λιθουανίας, τον κύριο Νάκος από τη Λιθουανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, οι τομεί ε, βιομηχανίας και γεωργίας σε ορισμένες χώρες πλήττονται από τις ε, ανισότητες ε, σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστική θέση των αγροτών γιατί ας πούμε οι αγρότες στη Γαλλία, την Ισπανία και άλλες χώρες ζητούν περισσότερες Ευρωπαϊκέ επιχορηγήσεις. Ωστόσο, οι υπόλοιποι αγρότε, από άλλες χώρες δεν έχουν λάβει τα κονδύλια που του αναλογούν. Δυστυχώ, οι μικρές χώρες, ιδιαίτερα από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, βρίσκονται σε δυσμενή θέση. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους ε, στόχους που έχουν αναλυφθεί για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των ωφέλων της ανταγωνιστικότητας αυτής. Οι περαιτέρω εξελίξεις θα έχουν σημαντική επιρροή ε, στις εθνικές μας οικονομίες γιατί οι χώρες αυτές οι μικρές δεν θα μπορέσουν ποτέ να ανταγωνιστούν πραγματικά τις ε, χώρες με καλύτερη χρηματοδότηση. Ε, οι άνεργοι προσπαθούν, προσπαθώντας να βρουν μια θέση εργασίας, ε, φεύγουν από τις χώρες μας, αναζητώντας ε, δουλειά σε άλλα κράτη-μέλη. Κατά αυτόν τον τρόπο, Ευρωπαίοι πολίτες από τη Λιθουανία και άλλες χώρες θα αναγκαστούν να ψάξουν δουλειά στα ναυπηγεία του Αμβούργου και αλλού. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συστήσουμε και άλλα μέτρα. Θα πρέπει να εστιάσουμε στην καλύτερη προστασία των εξωτερικών μας ενόρων. Πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας σε αυτό το τομέα, να καταπολεμήσουμε ε, το λαθρεμπόριο, ε, ιδιαίτερα μέσω και την εμπορία ανθρώπων, ιδιαίτερα διαμέσω της ε, Λευκορωσίας για να αυξήσουμε το ανταγωνιστικό μας ε, πλεονέκτημα στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ενισχύσουμε τις οικονομικές μας σχέσεις με τρίτες χώρες. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας ε, που θεωρώ ότι θα επηρεάσει ιδιαίτερα την ε, θετική εξέλιξη αυτού του θέματος. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο εκπρόσωπος του Γαλλικού Κοινοβουλίου. Ναι, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αυτή η πράξη για την αγορά θέλει να θέσει στο κέντρο αυτό και να τους, μας βάλει σε μια ανταγωνιστική αγορά. Εμείς σαν Γάλλοι το υποστηρίζουμε με την κοινωνική διάσταση της εταιρικής αγοράς και χαιρόμαστε για αυτή την ανάληψη που από την Επιτροπή να αναλύει αυτή την κοινωνική επίδραση όλων των νομοθεσιών στην εννέα αγορά. Και ιδιαίτερα υπερασπιζόμαστε την ανάγκη να εκτιμήσουμε αυτέ την, ε, αυτές τις ρυθμίσεις ε, τις ευρωπαϊκές. Και εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια λεπτότερη ανάλυση, λεπτομέστερη ανάλυση για αυτές τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις και σε επίπεδο κρατών μελών Λοιπόν. Γι' αυτό ακριβώ η προετοιμασία αυτών των ε, μελετών επιπτώσεων ε, είναι από τα κράτη-μέλη για να βελτιώσουν τι αναλύσει του για το πώ επέρνουν τα πράγματα στη χώρα τη δική του και ξεκινώντα ήδη στη σύνταξη των κειμένων και η Γαλλία ακριβώ ε, θα παίξει το ρόλο τη και θα συμμετάσχει όπω πρέπει. Επίση υπάρχουν δυσκολίε παρακολούθηση τη εφαρμογή αυτών των προτάσεων στα διάφορα κράτη-μέλη. Μήπω θα έπρεπε να το σκεφτούμε αυτό το πράγμα για ίσω να υπάρξει μια μεικτή γραμματεία με το Συμβούλιο, με το Κοινοβούλιο και με τα Εθνικά Κοινοβούλια και έτσι για να δούμε ακριβώς από το ξεκίνημα ήδη τα διάφορα προβλήματα και που λιμνάζει η κατάσταση και να υιοθετηθούν όσο γίνεται νωρίτερα αυτές οι οδηγίες. Για τις οδηγίες αυτές ακριβώς αναφερόμενοι, αυτός ο ιδιαίτερος χαρακτήρας, ο συγκεκριμένος χαρακτήρας των ειδηγιών δεν αφήνει ιδιαίτερο περιθώριο λιγμού στα κράτη-μέλη. Άρα λοιπόν η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο είναι κάπως δύσκολη. Μήπως θα πρέπει να έχουμε μια κάποια απλούστευση στον επίπεδο αυτό αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Έμμα Μακλάρκεν, μέλος του Ευρωκοινοβουλίου. Thank you. Um, I'd like to thank Madam... Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γαλενέση και όλου του συναδέλφου για τα σημεία που έχουν θίξει, ιδιαίτερα όσα είπαν κατά του προστατευτισμού και, τη, και, την, και τις ανάγκες μας ε, να εστιάσουμε στην βελτίωση της ε, ε, λειτουργίας της ε, ενιαίας αγοράς που είναι κύρια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα, ε, την, να αυξήσουμε τις θέσεις εργασίας αλλά να τονώσουμε και την καινοτομία. Ε, με βάση και την έκθεση που λάβαμε στην αρχή του ε, χρόνου μπορούμε να συμπεράνουμε ότι θα πρέπει βεβαίως να υπάρχει και μια κατάλληλη διαδικασία εποπτείας. Και ε, η ενιαία αγορά που έχει προτεθεί το 2009 είναι το κατάλληλο εργαλείο για να επιτευχθεί αυτό και για να διασφαλίσουμε ότι γίνεται η σωστή μεταφορά της νομοθεσίας. Μια άλλη πρόταση είναι η εναλλακτική επίλυση διαφορών. Εγώ χαιρετίζω αυτή την προσπάθεια. Είναι μια σωστή πρακτική που θα έχει προσταθέμενη αξία για του Ευρωπαίου πολίτε. Το θέμα για την. Ε, Πράγματι βρισκόμαστε σε ελιμνάζοντα νερά σε ότι αφορά την αύξηση του ανταγωνισμού και ε, κινδυνεύουμε να χάσουμε το παιχνίδι σε σχέση με άλλες χώρες, αναδυόμενες δυνάμεις όπως η Ινδία κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκλειδώσουμε, αν θέλετε, τα ωφέλη της ενιαίας αγοράς. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ένα κυβερνητικό έγγραφο που ε, καθορίζει πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό με την άρση των εμποδίων εμπορίου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, μείωση ε, του κόστους δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και προωθώντας την ψηφιακή επανάσταση. Σε αυτούς τους τομείς λοιπόν είναι πολύ σημαντική η οικονομική διακυβέρνηση στην αγορά. Και αυτή η καθοδήγηση των εισαγωγικών ε, είναι πολύ σημαντική για την ενιαία αγορά. Οι οδηγίες αυτές λοιπόν οι ευρωπαϊκές θα πρέπει να μεταφερθούν ε, εν ευθέτω χρόνο στις εθνικές νομοθεσίες. Ε, και βεβαίω θα πρέπει να ενημερωθούν και οι εταιρείε για το πώς το ευρωπαϊκό δίκαιο επηρεάζει την εθνική νομοθεσία προκειμένου πάντα να αρθούν και τα εμπόδια στο πλαίσιο των κρατών μελών. Η Επιτροπή, από την άλλη, θα πρέπει να συμβάλλει και αυτή με τη, τη μεριά τη σε αυτή τη διαδικασία. Η εταιρική σχέση ε, που ε, έχει δρεώσει με τα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να ενισχυθεί, προκειμένου να συνάψει ή μάλλον να διεξαγαγεί και διαπραγματεύσει εμπορικέ ε, με τα ενδιαφερόμενα μέρη στα κράτη-μέλη. Γιατί βεβαίως δεν πρόκειται για εύκολο καθήκον. Είναι μια μεγάλη πρόκληση αυτή, να καταφέρουμε να επιτύχουμε αυτή την ευημερία και την καινοτομία για να ε, προωθήσουμε την ε, ευρωπαϊκή μας οικονομία. Ευχαριστώ. Κυρία Μακλάρκεν. Ο κύριος Αντώνιο Κορέα Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω τρία πράγματα σύντομα. Πρώτα απ' όλα για την ε, ενσωμάτωση της ε, νομοθεσίας και τι ρόλο μπορεί να παίξει το θέμα αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να προσέξουμε πώς ακριβώς ε, όλα αυτά θα ενσωματωθούν και για τον αριθμό των οδηγιών, αλλά και για το περιεχόμενό τους αυτό καθ' αυτό. Άρα λοιπόν ε, στις κυβερνήσεις, στα κράτη-μέλη θα πρέπει να ανακοινωθούν και ενδεχόμενες καθυστερήσεις. Αυτό το είπα και στη δική μου την κυβέρνηση, δηλαδή σημείωσα τις καθυστερήσεις που σημειώνονται και δεν θα πρέπει να έχουμε και προβλήματα από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας. Θα πρέπει νομίζω να προσπαθούμε όλοι για θετικά αποτελέσματα. Τώρα για ορισμένε νομοθετικές διαδικασίες που προωθούν τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτή η διαδικασία δεν θα πρέπει να είναι μονομερής. Κανείς ε, δεν απαιτεί να διδάξει στους άλλους πώς θα πετύχουμε τη σύγκληση των διαφόρων νομοθεσιών, αλλά θα πρέπει να υποφεληθούμε από τις συναντήσεις μας και με το παράδειγμα της καλής πρακτικής και θα ήθελα να φέρω ακριβώς και το φόρουμ της Κρακοβίας, αλλά και στην Ουγγρική Προεδρία είχαμε συναντήσεις μεταξύ κοινοβουλευτικών επιτροπών που ασχολούνται με Αγορά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιτροπές ακριβώς κοινοβουλευτικών που ασχολούνται και με τον ανταγωνισμό, όπως ακριβώς και με μια επιτροπή από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Θυμάμαι ότι χρειάζονται προσπάθειες όχι μόνο από πλευράς Κοινοβουλίου. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ όταν μας έδωσε μια εικόνα σχετικά με τα μέτρα που αφορούν την ενία αγορά, οργάνωσε συναντήσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια σε όλες τις χώρες και ακριβώς ήθελα και θέλαμε όλοι μας να συμμετάσχουμε εκεί δυστυχώς οι εργασίες μας, τα καθήκοντά μας δεν μας το επιτρέπουν πάντα αυτές οι κοινέ συναντήσεις θα πρέπει να αφορούν και άλλους τομείς όχι μόνο την εσωτερική αγορά σίγουρα θα το καταφέρουμε αυτό και θα πρέπει να αποφύγουμε να λοκατηγορούμεθα θα πρέπει πρέπει να ξεχάσουμε, να βάλουμε στην άκρη, να βάλουμε σε παρένθεση και το θέμα του προστατευτισμού. Γιατί σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τι προσπαθούμε, να διδαχτούμε ακόμα πράγματα σχετικά με τις διευρυμένες αρμοδιότητες που μας αποδόθηκαν. Εδώ και δύο χρόνια το βλέπουμε αυτό. Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα. Τι παρατηρώ όμως, σε κάθε επίπεδο, σε κάθε κοινοβουλευτικό όργανο, Παντού συμμεριζόμαστε αυτές τις απόψεις και αν το συνεχίσουμε θα είναι θετικό για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Μίλλερ από την Ουγγαρία. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ακούσαμε ήδη ορισμένες λέξεις κλειδιά διαφάνεια, πληροφόρηση, ενημέρωση, διακυβέρνηση, συνεργασία, σε όλα αυτά συμφωνούμε. Εάν θέλουμε να εργαστούμε σωστά, πρέπει να εργαστούμε μαζί. Ε, συνεργασία λοιπόν. Άλλη, είναι μια λέξη κλειδί, μια έννοια κλειδί και ενημέρωση, αλληλοενημέρωση. Εχτες συζητήσαμε τις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές και την αξία της πληροφορίας. Ξέρουμε ότι πολλές, πολλοί πολίτες μας δεν έχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται διότι το σύστημα είναι αδιαφανές. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να το έχουμε στο, στην ατζέντα μας, στην ημερήσια διάταξη. Επίσης, το θέμα της παιδείας, διαμέσου δηλαδή της παιδείας, να ενισχυθεί η πληροφόρηση, η κατανόηση όλων αυτών των διαδικασιών που έχουν επίπτωση στη ζωή τους. Εάν δεν τους παράσχουμε την αναγκαία πληροφόρηση, οι πολίτες θα έχουν το αίσθημα ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω τους ε, είναι εντελώς ξένα, ακατανόητα πράγματα, στα οποία δεν έχουν καμία συμμετοχή και καμία επιρροή. Ο τύπος. Ο τύπος επίσης μπορεί να παίξει έναν σημαντικό ρόλο, έναν ενεργό ρόλο. Είναι πολύ σημαντικός ε, ο τύπος γενικά στην πληροφόρηση, στην ενημέρωση, έτσι ώστε οι πολίτες να καταλάβουν, να κατέχουν δηλαδή την ε, διαδικασία λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες. Ε, εάν οι πολίτες μας έχουν τις αναγκαίες πληροφορίες, θα συμμετάσχουν και πιο πρόθυμα. Είναι σωστό ότι ορισμένα κράτη-μέλη κάνουν μια έντονη προσπάθεια για να ενσωματώσουν περισσότερο τους πολίτες στη λήψη των αποφάσεων. Όμως, χρειαζόμαστε και θεσμικές διαδικασίες διαδικασίες οι οποίες θα αγκαλιάσουν τους πολίτες και θα τους φέρουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν αυτές οι πληροφορίες, αυτή η ενημέρωση δεν παρασχεθεί, εάν ε, οι διαδικασίες είναι κατανόητες και αδιαφανείς προς τους πολίτες, εάν οι πολίτες δεν παίξουν κανένα ρόλο στη λήψη των αποφάσεων, τότε αργά ή γρήγορα θα δημιουργηθούν οξύτερα προβλήματα και θα αναγκαστούν οι κυβερνήσεις να λάβουν προστατευτικά μέτρα. Και οποιοδήποτε μορφή προστατευτισμού δεν είναι θετικό μέτρο σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Ξέρουμε ότι υπάρχει και έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, γι' αυτό οι πληροφορίες πρέπει να, να ρέουν απρόσκοπτα και εδώ αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που αναφέρατε αυτή τη σημαντική πτυχή της διακυβέρνησης. Και τώρα θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Θα ήθελα να καλέσω την κυρία Καλιάτε να ολοκληρώσει τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Όχι, Ευχαριστώ ε, ιδιαίτερα για όλες ε, τις ε, παρεμβάσεις που έγιναν από το συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτή η συζήτηση έδειξε την παρουσίαση της σημερινή κατάσταση της ενιαίας αγοράς. Πολλοί ομιλητέ τόνισαν τη σημασία του διαλόγου μεταξύ Βρυξελών και Εθνικών Κοινοβουλίων. Στην έκθεσή μου για τη διακυβέρνηση και την εταιρική συμμετοχή διέθεσα αρκετές παραγράφους ε, στο θέμα του διαλόγου. Πράγματι, ε, κάθε δεύτερη παράγραφος μου έχει ε, κάποια αναφορά στο διάλογο μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ πολιτών και θεσμικών οργάνων της Ένωσης, μεταξύ ε, της, ε, ανάγκης διάδοσης ε, των πληροφοριών και της ανάγκης ενημέρωσης των πολιτών. Το, πώς θα γίνεται αυτή η ενημέρωση. Αλλά επανέρχομαι σε αυτά που είπε ο εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας. Είναι σωστά αυτά που είπε, διότι όλες αυτές οι ευρωπαϊκές αποφάσεις yes, λαμβάνονται από κοινού. Μαζί παίρνουμε τις αποφάσεις. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι μόνο υπεύθυνα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να παρουσιάσουν και να εξηγήσουν και να κάνουν κατανοητές τις αποφάσεις αυτές τους ε, Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και τα εθνικά κοινοβούλια έχουν ίση ευθύνη. Και τώρα αναφέρουμε σε ένα στοιχείο το οποίο αναφέρθηκε σε όλες τις παρεμβάσεις το πόσο περίπλοκο είναι το θέμα αυτό της ε, διακυβέρνησης και πόσο καλύτερα πρέπει να ε, είναι να χρησιμοποιούμε κανονισμούς. Ε, υπάρχει σαφώς μια μεγάλη περιπλοκότητα στα θεσμικά και νομοθετικά αυτά πλαίσια. Γι' αυτό ακριβώς και ζητάμε τη δημιουργία αυτών των πινάκων συσχετισμών των νομοθεσιών αυτό που θέλουμε είναι να μπορούν να μεταφέρονται και να εφαρμόζονται τα νομοθετικά μέτρα καλύτερα και ταχύτερα. Ο εκπρόσωπος της Σουηδίας τόνισε ε, τη σημασία του να μην επιβάλλουμε κάτι από την κορυφή προς τη βάση. Ε, δεν μπορούμε να διατάσουμε και να επιβάλλουμε. Όλα θα πρέπει να αποφασίζονται μετά από διάλογο, ακριβώς όπως τα κάνει η Επιτροπή μας, ΙΜΚΟ. Εμείς ε, αναμένουμε την συμμετοχή, την ε, παρέμβασή σας, το διάλογο σας, βασιζόμαστε στη συνεργασία σας. Επί χρόνια ήμουνα και εγώ εθνική βουλευτής και δεν έχω την εμπειρία αυτή της, της συνδιαλλαγής και του διαλόγου. Πιστεύω ότι την επόμενη φορά θα έχουμε ε, και άλλα θέματα να συζητήσουμε και σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κανιάντα για αυτή την εξαιρετική σύνοψη. Θα το κλείσουμε εδώ λοιπόν αυτό το θέμα της μέσης διάταξης. Παραδίδω και πάλι την Προεδρία στον ε, συνάδελφο. Τον κύριο Αντρέη Τρεβίνσκι από την Πολωνία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το επόμενο θέμα είναι εξίσου ενδιαφέρον, μια συζήτηση για την ε, ψηφιακή ενιαία αγορά, τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη, για τα κράτη-μέλη και για τον κόσμο. Ίσως ε, να το ξέρετε, αλλά είναι σημαντικό να θέσουμε και ένα πλαίσιο για να καταλήξουμε ε, σε επικοδοματικά συμπεράσματα. Η συζήτηση αυτή θα διεξαχθεί όπως και προηγούμενη ε, υπάρχουν ήδη ορισμένοι από εσά που έχουν ζητήσει το λόγο. Αν υπάρχει κάποιο διαδικαστικό ερώτημα, μπορείτε να το θέσετε τώρα. Όχι, εντάξει. Όπως και πριν. Θα γίνει και αυτή η συζήτηση. Αρχικά, Αντώνη Μέντζεβο, εκπρόσωπος της Πολωνικής ε, Γερουσίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ε, η οικονομική κρίση που έχει επιλέξει την Ευρώπη είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να συζητήσουμε το μέλλον της ε, ενιαίας αγοράς. Πέρσι εγκρίθηκε η στρατηγική για το 2020 για την Ευρωπαϊκή Ένωση που προσδιορίζεται και ο τρόπος ανάπτυξης της Ευρώπης. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ είπε ότι η ενιαία αγορά είναι κλειδί για ε, την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και η, η επαναφορά αυτή στην ε, πρόοδο και την ανάπτυξη απαιτεί προσπάθειες ε, για την καταπολέμηση της κρίσης τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό βεβαίω, όσο και σε παγκόσμιο θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να πετύχουμε μια ψηφιακή ενιαία αγορά στην Ευρώπη και η ευρωπαϊκή αγορά είναι διατεθειμένη να αναλάβει αυτό το καθήκον για να βρεθεί σε καλύτερη ενταγωνιστική θέση. Αυτό πρέπει να γίνει με γρήγορη ε, προσαρμογή στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Αγαπητά μέλη των κοινοβουλίων, αυτή η δημιουργία της ε, ψηφιακή εσωτερικής αγοράς είναι μια τεράστια πρόκληση για τους πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικονομία δεν είναι έτοιμη για τον παγκόσμιο ανταγωνισμό ε, και δεν θα είναι έτοιμη έως ότου ε, γίνουμε πιο ανοιχτοί στην ψηφιακή αγορά. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι τομείς θα πρέπει να λάβουν ιδιαίτερη στήριξη τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Πρώτον, η εσωτερική αγορά θα πρέπει ε, να καλύπτει τις ε, φιλοδοξίες και τις ανάγκες νέων επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ολοκληρωμένη αυτή η αγορά χωρίς εμπόδια. Και τρίτον, θα πρέπει να, παρέχουμε στήριξη και στον ε, τομέα του εμπορίου προσπάθειε θα πρέπει να καταβληθούν στον τομέα των υποδομών ε, ε, τη ψηφιακή τεχνολογία, Ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το στοιχείο, ε, συνιστόσα τη κοινωνίας τη πληροφορία. Και θεωρώ ότι στο μέλλον δεν θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια κοινωνία της πληροφόρησης αν δεν αξιοποιήσουμε και όλες αυτές τις τεχνικές δυνατότητες που μας παρέχει. Τώρα για να φτάσουμε να καταλήξουμε σε μια τέτοια ψηφιακή ενιαία αγορά ε, μπορούμε να διαβάσουμε και το κείμενο της Επιτροπής, την ανακοίνωση για τη στρατηγική 2020. Εκεί βλέπουμε και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το με αυτό. Εφτά ε, προγράμματα αναφέρονται εκεί. Ένα από αυτά είναι το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Θυματολόγιο, European Digital Agenda, η παροχή μιλά για, την, ε, ε, για τους παρόχους ε, διαδικτύου και, και εκεί πέρα αναφέρεται ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές από χώρα σε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά την ψηφιακή αγορά. Γι' αυτό η Επιτροπή θέλει να αναλάβει δράσεις προκειμένου να υπάρχει μία και ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην οποία θα έχουν εύκολη πρόσβαση οι πολίτες. Οι συναλλαγές μας του διαδικτύου να καταστούν πιο εύκολες προκειμένου οι Ευρωπαίοι πολίτες να δουν πόσο ελκυστική είναι μια τέτοια αγορά, πόσες ε, περισσότερες επιλογές τους ε, δίνει ε, για παράδειγμα, το να έχουν μια ε, αξιόπιστη και έναν αξιόπιστη και εύκολο τρόπο πληρωμών μέσω διαδικτύου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να, υπάρχει και σωστέ, να υπάρχουν σωστές ρυθμίσεις για την προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων. Αλλά και οι τηλεπικοινωνίες και οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα πρέπει να προσαρμοστούν καταλήλως. Σε αυτό το έγγραφο βλέπουμε αρκετές ε, πρωτοβουλίες και ενέργειες. Μία από αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ε, αυτό το ψηφιακό θεματολόγιο. Εμεί στηρίζουμε όλες ε, αυτές τις προτάσεις. Η Επιτροπή αναφέρει την ύπαρξη εμποδίων, για παράδειγμα ο κατακραματισμός της αγοράς την έλλειψη προστασίας ή μάλλον την ελλειπή ε, προστασίας ε, ελλειπή προστασία των καταναλωτών στην ψηφιακή αγορά. Και ουσιαστικά βλέπουμε ότι παραμένουν δυσκολίες ε, στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Και αυτό είναι κρίμα. Βλέπω ότι δεν έχω αρκετό χρόνο. Απλώς θέλω να αναφέρω τα, ότι υπάρχει μεγάλο όφελος ε, ε, στην ε, σωστή και ομαλή λειτουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Μας προσφέρει πιο εύκολη πρόσβαση στην καινοτομία, μεγαλύτερη ευκολία στη λειτουργία των μικρών και μεσών επιχειρήσεων αλλά προωθεί και την οικονομική ανάπτυξη στο σύνολό της και βεβαίω τεράστια ωφέλη για τους καταναλωτέ. Ιδιαίτερα ε, σε ό,τι αφορά υπηρεσίες ε, και αγαθά και, την, και τις στο διαδίκτυο. Σημαντικά είναι το ωφέλη και για τις διοικήσει, για τα κράτη. Μπορεί να λειτουργούν, έχουν δυνατόν να λειτουργούν καλύτερα και πιο σωστά και ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίση, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν καταφέρουμε μέχρι το 2020 να καταλήξουμε στην ομαλή, να επιτύχουμε μάλλον την ομαλή λειτουργία της ψηφιακής αγοράς, θα έχουμε τεράστια πρόοδο. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, ιδίω για αυτή την αισιόδοξη ε, εισαγωγή σας. Ο κύριος Ντεκάμπος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά Λάουρα ε, Γαλλία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον συνάδελφο Αντιπρόεδρο του Πολωνικού Κοινοβουλίου για την άριστη παρουσίασή του. Σίγουρα ήταν αισιόδοξο όπως είπε και ο Πρόεδρος αλλά μας έδειξε ταυτόχρονα χαράσοντάς μας τις κατευθύνσεις για το μέλλον. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο οι τάσεις είναι ότι έχουμε ακόμα 9% διαμεθοριακό εμπόριο παρόμοιο και όταν κάνουμε μια διάγνωση της καταστάσεως συμφωνούμε ότι χρειάζεται ένα διατραπεζικό, πιο ρευστό, πιο ευέλικτο σύστημα που να εμπνέει εμπιστοσύνη, επίσης ένα κατάλληλο φορολογικό σύστημα και ένα καλό ταχυδρομικό σύστημα ώστε να μπορούν τα πράγματα να παίρνουν μια μεριά στην άλλη και πολλές και διάφορες πτυχές που έχουν να κάνουν επίσης με πολιτιστικά σημεία οι ψηφιακές προκηρύξεις ε, διαγωνισμών και προσκλήσεις ενδιαφέροντος μπορούν να εξυπηρετήσουν για αγορές του δημοσίου, θα μπορεί να είναι κάτι το πολύ θετικό για να δώσουν μια όθηση σε αυτό το εμπόριο, γιατί μας υποχρεώνουν σε μια τυποποίηση, σε μια πειθαρχία, στη δημιουργία ε, εργαλείων τραπεζικών και επίσης χρησιμοποιούν και τον ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα χρειάζεται να υπάρχει εμπιστοσύνη. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη για τις τεχνολογίες. Οι πλατφόρμες που δουλεύουν καλύτερα σε αυτό το εμπόριο βασίζονται στην εμπιστοσύνη από οικονομικής πλευράς και επίσης για την ε, privacy και μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή που προώθησαν ιδιαίτερη δραστηριότητα στον τομέα αυτό. Είμαστε σε θέση να συστήσουμε ένα μόνιμο παρατηρητήριο του ηλεκτρονικού εμπειρίου για να ενημερωνόμεθα για τις καθυστερήσεις μας και γνωρίζουμε ότι ναι, έχει σημειωθεί ιδιαίτερη καθυστέρηση και θα πρέπει πολλά να γίνουν γύρω από αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι, πράγματι, η εμπιστοσύνη στον τομέα του εμπορίου είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και σίγουρα όλες αυτές οι τακτικές ε, παραβιάσεις του κυβερνοχώρου από τους λεγόμενους hackers <clears throat> δεν βοηθούν την κατάσταση. Θα δώσω τώρα το λόγο στον, στη Λάγα από τη Γαλλία. Και μετά, Όλε Johansson. Ε, Σας ευχαριστώ θα βασιστώ σε ορισμένα σημεία επίκαιρα σε εθνικό επίπεδο στη Γαλλία που ανησυχούν γενικά την Ευρώπη και θα πρέπει να δούμε την πραγματικά το ίντερνετ είναι από τους φορείς ανάπτυξης ε, παρόμοιας ψηφιακής δραστηριότητας ε, και που είναι επικερδής σε όλους κυρίως εκείνους που ασχολούνται με το περιεχόμενο και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε. Μετά από το τρίτο ε, δέσμι Telecom όμως αυτοί οι δέσμοι είναι ανεπαρκείς. Δεν έχουν υπάρξουν, ε, δεν υπάρχουν ε, απέναντι σε σημαντικούς φορείς παροχή υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, θεωρούμε ότι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η θέση στην ανακοίνωση του Απριλίου 2011 είναι κάπως άτολμη και θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να παρατήσετε από κοντά την εργασία του Εθνικού Κοινοβουλίου σχετικά με την ουδετερότητα αυτή του ίντερνετ. Δεύτερο, νέα δίκτυα νέας γενιάς για τις οπτικές ίνες μέσω αυτών και παρόμοια δίκτυα οπτικών ινών αποτελεί πρόκληση ιδιαίτερα για την οικονομία αυτή σε επίπεδο Ευρώπης και χρηματοδότηση για αυτές τις οπτικές ίνες είναι 26 δισεκατομμύρια ευρώ αλλά δεν χρηματοδοτείται από τους ιδιωτικούς φορείς είτε από το δημόσιο. Γι' αυτό λοιπόν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είδαμε την πρόταση του Λίκρος Ευρωπαϊκό η για τη μείωση του φόρου πάνω σε αυτά εκτός αν θέλουν ακριβώς να επενδύσουν στις οπτικές σύνες. Και επίσης κάτι άλλο. Αναρωτιόμαστε για την ε, ε, πλατιά κάλυψη στο επίπεδο 2013, όπως την προωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί εκφράζουμε διάφορες αμφιβολίες για την κατάλληλη αυτή η στόχη, γιατί η περισσότερη ροή ίσως καθυστερήσει τελικά τη χρησιμοποίηση των οπτικών ινών, που σας επαναλαμβάνω ότι υποτέχει μια ιδιαίτερη πρόκληση για την ανάπτυξη αυτής της, του είδους της οικονομίας. Επίσης η Ευρωπαϊκή Στρατογική επιμένει και είναι καλό αυτό για τις υπηρεσίες, για το περιεχόμενο, για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και όπως και ο προηγούμενος ομιλητής θα επιμείνουμε στο ότι χρειάζεται φορολογικό συντονισμό σε κοινοτικό επίπεδο. Απόλυτα απαραίτητο είναι για να μπορέσει να αναπτυχθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επίσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέλαμε να προσκαλέσουμε να δειχτεί ιδιαίτερα φιλόδοξη σε αυτό το τομέα και διάφορες χώρες άλλωστε, πολλά κράτη-μέλη έχουν κατανοήσει τι ακριβώς αποτελεί σαν πρόκληση για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι, πράγματι χωρίς υποδομές ε, δεν πάμε μακριά. Αυτό είναι σαφές. Και γι' αυτό είναι προφανώς ότι εκεί θα πρέπει να γίνουν οι επενδύσεις. Όλοι Γιώχανσον. Ευχαριστώ. Ε, η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών σημείωσε ότι η Σουηδία και η Νότια Κορέα είναι ε, δύο από τις πιο αναπτυγμένες χώρες ό,τι αφορά αυτόν τον τομέα. Πολλοί Σουηδοί πολίτες έχουν ίντερνετ στο σπίτι, όχι όλοι βεβαίως. Ε, αρκετοί έχουν και μάλιστα σύνδεση υψηλή ταχύτητα, όχι όλοι όμως. Ε, παρέχουμε υπολογιστές σε μαθητές, αλλά σε, όχι σε όλους. Και πολλοί πολίτε χρησιμοποιούν ε, τους του τους ε, για τις ε, τραπεζικές συναλλαγές και το καθεξής, αλλά όχι όλοι και πάλι. Ε, πολλά είναι τα εμπόδια μείωση κινητικότητα, ε, ηλικία, διάφοροι άλλοι παράγοντε για την ψηφιακή περιθωριοποίηση αν θέλετε. Αυτά λοιπόν τα εμπόδια θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικές γενιές ε, θα έχουν σίγουρα πρόσβαση στην ψηφιακή ενιαία αγορά όλοι δηλαδή να έχουν αυτή την πρόσβαση στο μέλλον. Θεωρώ ότι ο τομέας της πληροφορικής ε, θα μας βοηθήσει ε, και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ε, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, και στην καλύτερη αξιοποίηση και διαχείριση των φυσικών μας πόρων. Ο πληθυσμός μας σίγουρα γερνά, αλλά είναι και πιο μορφωμένος, πιο ενεργός, ξέρει πώς να αξιοποιήσει τα εργαλεία πληροφορικής και αυτό θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε το βιωτικό επίπεδο, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένου. και πρέπει να εξετάσουμε και τις προοπτικές της, ε, του τομέα της πληροφορικής ε, στον τομέα της ε, υγείας, στην διεξαγωγή χειρουργείων και ούτω καθεξής προκειμένου να βρούμε την καλύτερη και βέλτιστη ε, θεραπεία για κάθε πολίτη. Τέλος, ε, τα κοινωνικά μέσα επικοινωνίας ε, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την επικοινωνία των πολιτών διασυνοριακά, αλλά βεβαίως αυτό επιτρέπει και την ύπαρξη διαφορετικών απόψεων και την ανταλλαγή τους. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ε, την ε, ανοιχτή λειτουργία ε, αυτών των εργαλείων διεθνώς. Μπορούμε να δούμε τι έγινε στην Νότια Αφρική πρόσφατα και τι σημαίνει αυτό για την ελευθερία ε, και το δικαίωμα ε, ελεύθερης έκφρασης ε, των πολιτών. Επίσης, σε ό,τι αφορά το λεγόμενο roaming, την περιαγωγή και τις χρεώσεις, θα πρέπει να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού, γιατί βεβαίως όλοι έχουμε κινητά τηλέφωνα το δίκτυο τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να αναπτυχθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολίτες να είναι έτοιμοι να αξιοποιήσουν και αξιοποιήσουν την πληροφορική και στα σχολεία. Θα πρέπει τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια να έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τις ικανότητε του στον τομέα της πληροφορική. Πολύ σημαντική η παρέμβασή σα. Ούμπερτ Κούστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μπορούμε να τα επιβεβαιώσουμε όλα αυτά. Η εσωτερική ψηφιακή αγορά μας προσφέρει δυνατότητες αλλά ενέχει έχει και κινδύνους. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη όπως επίσης και η ασφάλεια, η προστασία των στοιχείων μια ασφάλεια απέναντι στο ε, έγκλημα στο διαδίκτυο. Είναι σημαντικά όλα αυτά για να μπορέσει να εξελιχθεί αυτή η αγορά θετικά. Χρειάζονται όμως ενιαίες οδηγίες ε, για τον τρόπο δράσης για την ασφάλεια, για τον καταναλωτή. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι πληρωμές μέσω του ίντερνετ θα φτάνουν στον αποδέκτη τους ακριβώς. Και χρειάζεται μία επαγρύπνηση για κατάλληλη επιλογή και θα πρέπει να υπάρξει το προϊόν που να προσφέρεται ποιοτικό και θα ήθελα να σας περεπέψω στο θέμα της πειρατείας που όλο και περισσότερο έντονο γίνεται αυτό και θα πρέπει να βελτιωθούν αυτές οι υπηρεσίες στο ίντερνετ χωρίς γραφειοδιακ ε, γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις και σε περίπτωση εγγύη, σε περίπτωση παραπώνων και διένεξης νομικής χρειάζεται να ισχύει αυτή η οδηγήση. Αυτό. να υπάρχει εξασφάλιση επίσης χρειάζεται να επιβλέψουμε, να προστατεύσουμε τα στοιχεία και τα εμπιστευτικά στοιχεία που δίδονται στις αρχές αποδεικνύουν ότι οι ιδιώτες ε, ή οι αρχές δεν αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό και χρειάζεται στον τομέα αυτό να προσπαθήσουμε και να επενδύσουμε. Και κάτι το τελευταίο τα παιχνίδια στο ίντερνετ. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, καμία ρύθμιση πάνω σε αυτό και θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει όσον αφορά τα κέρδη, τη φορολογία στα κέρδη, όλα αυτά χρειάζεται να ελέγχονται και υπάρχουν δυσκολίες όμως, ε, μάλλον παρατηρούνται δυσκολίες ε, και ανοίγουν καινούριε δυνατότητες για τους εγκληματίες. Χρειάζονται προσπάθειες και ψυχολογικές και πραγματικές. Τα παιδιά υποφέρουν από αυτό και υπάρχουν στην Αυστρία περιορισμένα παιχνίδια, τα πούμε έτσι, με καλύτερη ρύθμιση για τον περιορισμό της εγκληματικότητας. Αυτά θα ήθελα να πω σχετικά με το σημείο αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση. Πράγματι, ε, η εμπιστοσύνη του πολίτη και το αίσθημα ασφάλεια είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη τη αγορά. Να δώσω τώρα το λόγο στον πρόεδρό μα. Μόλκο Μουχάμπε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σε αυτήν την περίπτωση μιλάω και ως ε, μέλος της ομάδας, όσο και ως εισηγητής στην Επιτροπή για το πακέτο τηλεπικοινωνιών. Ε, ορισμένες γενικές παρατηρήσεις έχω να κάνω. Να σας δώσω μερικά στοιχεία για τους τομείς ε, στους οποίους εργαζόμαστε. Είναι ε, ε, τομέας κρίσιμης σημασίας για, τις, για την κοινή μας συνεργασία γιατί είναι ένας τομέας όπου θα πρέπει να επιτευχθεί πρόοδος σε κάθε χώρα. Η υπήρξε μια έκθεση της Επιτροπής που εκδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και ένα από τα ζητήματα στα οποία αναφέρεται είναι η συνεργασία μεταξύ των δημοσίων αρχών και των φορέων ε, τυχερών παιχνιδιών. Γενικά θα ήθελα να αναφέρω ότι το Κοινοβούλιο στην άποψή του για το πακέτο των επικοινωνιών διαφώνησε με την αρχική ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα ε, και θεώρησε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στους εθνικούς φορείς. Το καλύτερο θα ήταν να υπάρχει μια κοινή συντονιστική δομή για να διασφαλιστεί ε, μια συντονισμένη εφαρμογή αυτό σε εθνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, η κυρία Τελαργογιά αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε, στο Νάσερ, σε έναν από τους καλύτερους ρυθμιστές. Σημαντικό αυτό το στοιχείο. Η κυρία Τελαργογιά νομίζω δεν με ακούει, αλλά εγώ απαντώ σε κάποια από τα ζητήματα που ανέφερε. Καλό θα ήταν να φορέσει τα ακουστικά της. Ε, μίλησε για ουδετερότητα του δικτύου. Η Επιτροπή θεωρεί πολύ ενδιαφέρον αυτό το σημείο. Υπάρχει και μια διαθέσιμη έκθεση που βεβαίω και μπορώ να σα στείλω. Ε, δεν συμφωνούμε με την Εθνική Βουλή της Γαλλίας αυτή τη στιγμή. Έχουμε δώσει στους ε, ρυθμιστές και ε, στους φορείς τη δυνατότητα να δράσουν από μόνοι τους. η ε, Υπάρχει λοιπόν θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις, ε, τις εξουσίες που ήδη διαθέτουν να θέλουν να παρέμβουν. Οι ρυθμιστέ θα δώσουν και τις δικές τους απόψει στα τέλη του χρόνου και θα δούμε τι έχουν να μας πούν και εκείνοι. Κλείνοντα, ε, συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία Ντελαγοντιέγα για τη σημασία των επενδύσεων. Και η κύρια πτυχή του αυτού του πακέτου τηλεπικοινωνιών είναι ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε άλλους επενδυτές ε, να επενδύσουν γιατί ακόμα έχουμε χώρες ε, που ακόμα ε, κυριεύονται αν θέλετε από τους παλιούς σχεδόν αρχαϊκούς προμηθευτές και παρόχους. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει και εμείς να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ευρεία πρόσβαση στο διαδίκτυο και ο στόχος των 30 ε, ε, μέχρι το 2013 δεν είναι υπερφιλόδοξος. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε. Και ήδη και σε αυτό το κτίριο βλέπετε ότι όσοι από εμά έχουν ε, iPad και iPhone, ε, ήδη έχουμε νέε λειτουργίε διαθέσιμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να δώσω το λόγο στην Άννα Μύρια Καρατσαβούλτ. Ευχαριστώ, συγγνώμη που καθυστέρησα, υπήρξε η καθυστέρηση στη μου. Πολλά θα έχουν υποθεί σίγουρα από του συναδέλφου μου, όμως ήθελα να αναφερθώ ε, στην σημασία της οικοδόμηση τη ψηφιακή Ευρώπη Σε μια εποχή που επιτέλους ε, κατανοούμε σιγά σιγά ότι ε, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στα, στις κρατικές επιχορηγήσεις για την αύξηση και την ανάπτυξη. Η ψηφιακή αγορά είναι σημαντικός πυλώνας για την πρόθεση της ανάπτυξης και της οικονομία και προφανώς υπάρχουν ορισμένα εμπόδια, περιορισμοί, ε, αγκυλώσεις που εμποδίζουν την παροχή υπηρεσιών στο διαδίκτυο και δεν αξιοποιούμε στο έπακρο τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Την προηγούμενη εβδομάδα ε, στην Πολωνία, έμαθα μάλλον ότι στην Πολωνία ε, την προηγούμενη εβδομάδα ε, υπήρξε δυνατότητα χρήσης του iTunes επιτέλους. Ε, επίσης έχουμε το πρόβλημα ότι σε, σε διαφορετικές χώρες υπάρχουν διαφορετικές τιμές για τα ίδια προϊόντα. προϊόντα. Ή σε ορισμένες χώρες ε, υπάρχουν προϊόντα που δεν είναι καν διαθέσιμα. Για παράδειγμα τα ιδιαίτερα αυτά ε, τα δικά γυαλιά 3D. είναι σημαντικό λοιπόν να προωθήσουμε πραγματικά αυτήν την ε, ψηφιακή αγορά, το διαδίκτυο είναι ένα μέσο. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει και πάλι εναρμόνιση, να υπάρχουν κοινοί κανόνες, ε, να αρθούν τα εμπόδια, αλλά και ε, να μειώσουμε το βάρος που θα πρέπει να επομιστούν οι επιχειρήσεις ο συνάδελφος ο Παύλο, ε, που είναι πραγματικά ο γκουρού σε ό,τι αφορά το εμπόριο στην Επιτροπή μας, θα έλθει σε λίγο. Αλλά ε, χαίρομαι που η Επιτροπή εστιάζει στον τομέα της πειρατείας και, του, ε, και της παραχάραξης προϊόντων. Είναι πολύ σημαντικός τομέας. Θέλουμε και αναμένουμε την οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές Προκειμένου να υπάρξει διαλειτουργικότητα, πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε στην ε, μείωση του κόστους περιαγωγής και ε, βριζονικό δίκτυο για όλους. Ελπίζω ε, μέτρα να ληφθούν και σε εθνικό επίπεδο για την άρση των υφισταμένων εμποδίων για να έχουμε μια ψηφιακή ευρωπαϊκή αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία τα είπατε. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Γκέμπαρτ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ που εσύ για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Πρόκειται για πολύ σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν τους πολίτες στη σημερινή εποχή δεν γίνεται να προχωρήσουμε χωρίς τα νέα αυτά επικοινωνιακά μέσα και γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Γιώχανσεν που είπε ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτό το τομέα για να μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Γι' αυτό πρέπει επίσης να φροντίσουμε την ευρυζωνική πρόσβαση για όλους και να θεωρηθεί ως καθολική υπηρεσία διότι πολλοί πολίτες δεν θα μπορέσουν να καλύψουν το κόστος της ευρωτιζωνικής σύνδεσης. Και άλλο ένα θέμα της πρόσβασης είναι η ουδετερότητα του δικτύου. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις ή πάροχοι να έχουν μια πλεονεκτική μεταχείριση ή πρόσβαση ε, στο δίκτυο έναντι των πολιτών. Ουδετερότητα λοιπόν. Πρέπει να φροντίσουμε να μην δημιουργηθούν διακρίσεις εναντίον των πολιτών. Αυτή η πολιτική της αποφυγής διακρίσεων είναι υψίστης σημασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτο σημείο είναι η προστασία δεδομένων, το οποίο αναφέρθηκε αρκετές φορές. Πολλοί πολίτες δεν προσέχουν δεν την ε, φύλαξη των προσωπικών τους, των ατομικών τους στοιχείων και έχουμε πλέον ε, την εμπειρία ε, και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δίκτυα υποκλοπής ε, τα οποία τα, τα, οποία χειρίζονται κακοποιά στοιχεία πολλές φορές τα οποία υποκλέπτουν ή κατασκοπεύουν τα ατομικά στοιχεία των πολιτών. Δεν μπορεί λοιπόν να ζητάμε διαφάνεια ε, στην πολιτική μας και ε, στην νομοθεσία μας, αλλά ταυτόχρονα να μην επιβληθεί διαφάνεια στην προστασία των δεδομένων των πολιτών. Προστασία λοιπόν των προσωπικών στοιχείων. Πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Όπως βλέπετε, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε στην Ένωση και στα ε, κράτη-μέλη. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω μερικά πράγματα για, τα ζητήματα πληροφορική. Ε, η Επιτροπή είπε ότι αν σε αυτή η ψηφιακή αγορά μπορούμε να σημειώσουμε τεράστια πρόοδο σε οικονομικά, από οικονομικής πλευράς βλέπουμε στο Κοινοβούλιο ακόμα λειτουργούμε με τα Windows 2003, το οποίο είναι σχεδόν 10 ετών και πάλι δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω από τα να στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εμένα μου φτάνει αυτό. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να έχουμε περισσότερα μέσα πληροφορική στη διάθεσή μα. Αυτό λέμε όταν ερχόμαστε εδώ, αλλά μετά όταν επαναρχόμαστε στι πρωτεύουσέ μα. Ε, τα κάνουμε όλα λίγο πιο ήπια. το βλέπουμε αυτό και με τα τυχερά παιχνίδια, με το online gambling. Ε, εμένα δεν με αφορά βέβαια προσωπικά γιατί εγώ δεν το κάνω αυτό. Ε, και άλλα μετά, ενώ όλοι λέμε ότι και συμφωνούμε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε αυτό το τομέα, στο τέλο δεν κάνουμε τίποτα. Πριν ε, δύο χρόνια, σα δώσω ένα παράδειγμα, συμμετείχα σε ένα πρόγραμμα για τα ε, βιντεοπαιχνίδια και δεν έχει σημειωθεί ούτε ένα βήμα. Και όταν βλέπω ότι στο, στις Ηνωμένες Πολιτείες το Kinect έχει γίνει σχεδόν εθνικό άθλημα ε, και έχει μπει ακόμα και στα σχολεία, αυτό με στενοχωρεί και με λυπεί γιατί βλέπω ότι όταν δεν γνωρίζεις κάτι, δεν κάνεις κάτι. Αυτό φαίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το, το οι πολίτες μας δεν το γνωρίζουν, οπότε λένε εντάξει δεν θα είναι και τίποτα τρομερό. Γι' αυτό, Πρόεδρε, θεωρώ ότι μπορούμε να ε, επιτύχουμε ε, αυτή την πρόοδο, να πάμε πραγματικά στα εθνικά μας κοινοβούλια και να τους ζητήσουμε να αναλάβουν μέτρα. Γιατί αν πραγματικά, αν πραγματικά μπορούμε να, ε, δημιουργήσουμε 900.000 θέσεις εργασία, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε με ευρωπαϊκό τρόπο νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε πολύ πιο δύσκολους από οικονομικής πλευράς καιρούς. Ε, Βεβαίω θα πρέπει να υπάρχει ουδετερότητα στο δίκτυο και όλα αυτά που αναφέρθηκαν. Βεβαίω να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να έχουμε το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον ε, και να άρουμε τα, τα σύνορα, αν θέλετε, και όλα αυτά τα εμπόδια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. η εθνική πολιτική, οι πολιτικοί μάλλον που προέρχονται από τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά και οι ευρωβουλευτές, θα πρέπει να ε, ακολουθήσουν τη στρατηγική για το 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας και που ήταν πολύ έντονη, με πολύ πάθος. Πολλοί από εμά χρησιμοποιούμε τη βελτιωμένη υποδομή, αλλά θέλουμε να εγγυηθούμε την ισότιμη πρόσβαση στις ε, τεχνολογίες σε όλους τους πολίτες. Η κυρία Έλτεγκάρτ από την, το Νορβηγικό Κοινοβούλιο. Ε, thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή και πολλά ενδιαφέροντα θέματα αναφέρθηκαν. Πιστεύω ότι οι πολιτικές που εφαρμόζουμε πρέπει να ανταποκρίνονται στους στόχους μιας πιο έξυπνης αηφόρου και ε, σωστής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Πάντως πρέπει να ξεπεράσουμε πολλά εμπόδια στην εσωτερική αγορά για να υποφεληθούμε της ψηφιακής αγοράς. Μια σωστά λειτουργούσα ε, ε, ψηφιακή αγορά μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν συνεργαστούν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να, να βρούμε ένα σύστημα διασυνοριακά για την ηλεκτρονική υπογραφή και τις ηλεκτρονικές επικυρώσεις. Επίσης, σύμφωνα με τον κύριο Γιώχανσον από τη Σουηδία, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να επωφεληθούν ισότιμα τις δυνατότητες της νέας ψηφιακής αγοράς. Ευχαριστώ. E, Ευχαριστώ. Υπάρχει ακόμα ο κύριος Ντεμικράν από το Τουρκικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ψηφιακή μετάδοση στοιχείων, δεδομένων γίνεται όλο και πιο σημαντική στις επικοινωνίες. Όμως η τιμολόγηση της κινητής τηλεφωνίας στα roaming είναι ακόμα υπερβολικά υψηλή ιδιαίτερα σε χώρες που είναι εκτός Ένωσης. Πιστεύω ότι αυτό το έχουν θίξει πάρα πολλές οργανώσεις καταναλωτών και ελπίζω να μπορέσει η Ένωση να μειώσει τις τιμές του Ρώμη και να προστατεύσει τα δεδομένα. Σύμφωνα με μία μελέτη του 2010, η Ένωση μπορούσε να κερδίσει 4% του ΑΕΠ μέσω της ανάπτυξης μέχρι το 2020 της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Αυτό ανταποκρίνεται σε 500 δις ευρώ. Όμως υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά εμπόδια τα οποία εμποδίζουν τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Όταν, αν ξεπεραστούν και όταν ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, τότε όλες οι οικονομίες πλέον θα λειτουργούν σε ψηφιακό επίπεδο. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ε, παρουσιάσω μερικές πληροφορίες, ορισμένα στοιχεία και σας ζητώ να προσέξετε το, το, το γεγονός ότι η πλήρης ένταξη της Τουρκίας δεν θα ωφελήσει μόνο την ε, Τουρκία αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία έχει μια αναπτυσσόμενη οικονομία και η ενσωμάτωση της τουρκικής οικονομίας στην ενιαία αγορά θα ωφελήσει και τις δύο πλευρές η, επίσης, το να γίνει μέλος η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι έτσι θα μπορέσουν οι ευρωπαϊκές αρχές της, δημοκρα... της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης να επεκταθούν μέσω Τουρκίας και πέραν από τη λεκάνη της Μεσογείου. Γι' αυτό πιστεύω εν συντομία ότι η πλήρης ένταξη της Τουρκίας δεν θα αποτελέσει βάρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά θα αποτελέσει όφελος. Γι' αυτό θέλουμε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις οι οποίες δυστυχώς έχουν κολλήσει και τα 18 κεφάλαια, κεφάλαια των διαπραγματεύσεων έχουν κολλήσει λόγω απλών πολιτικών ε, ε, αιτίων. Γι' αυτό θέλει το Κοινοβούλιο, θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πιέσει να υιοθετηθεί το κοινοτικό κεκτομένο ε, στις ε, διαδικασίες ένταξης της Τουρκίας. Όχι μόνο θέλουμε να γίνουμε πλήρες μέλος, αλλά πιστεύουμε στις ευρωπαϊκές αξίες και πιστεύουμε ότι ε, οι αξίες που προέρχονται από την Ευρώπη είναι αποτέλεσμα του ενιαίο ευρωπαϊκού πνεύματος. Γι' αυτό δεν θέλουμε να κολλήσει η ένταξή μας σε, πολιτικές, σε πολιτικά αίτια, λόγω πολιτικών αιτίων και τεχνικών προσκομμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Το ερώτημα είναι εάν η Τουρκία θέλει να ενταχθεί που θέλει και αν οι Ευρωπαίοι τι θέλουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Τούρκο συνάδελφό μας και σας εύχομαι δύναμη και επιμονή ε, στην, ε, στον αγώνα σας για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μπορεί επίσης και λάβουν μέρος στη συζήτηση, όπως ε, είπε και ο πρόεδρος μας εξ αρχής, ε, ε, τα παρευρισκόμενα μέλη εδώ στην αίθουσα, αν θέλετε, μπορείτε να σηκώσετε την μπλε κάρτα σας. Ο κύριος Βαλκιώνας έχει ζητήσει το λόγο, εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου της Λιθουανίας. Ευχαριστώ. όλοι ξέρουμε, βλέπουμε ότι ζούμε σε έναν παράδοξο κόσμο. Εχθές στην αίθουσα είχαμε καφέ, νερό, ε, ενώ σήμερα δεν έχουμε ούτε μία σταγόνα νερού να πιούμε. Αυτά εισαγωγικά. Λοιπόν, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και σύγχρονη τεχνολογία, όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Πρέπει όμως να προσφέρουμε καλύτερες τιμές, μεγαλύτερα ωφέλη στις επιχειρήσεις, περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές μας ε, σε, μια σωστή διάσταση κόστους ωφέλους. Αλλιώς πώς θα αλλάξουμε τις κοινωνίες. Πώς θα βρούμε λύσεις στην αυξανόμενη ανεργία πώς θα ε, χαλιναγωγήσουμε το αυξανόμενο κοινωνικό κόστος. Μπορεί το ηλεκτρονικό εμπόριο, ας πούμε, να συνδέεται και με ανεπιθύμητες επιπτώσεις, ξέρω εγώ, φοροδιαφυγή, ε, επιπτώσεις τις οποίες δεν θέλουμε, αρνητικές επιπτώσεις. Τι θα κάνουμε επίσης για την πιο εύκολη κυκλοφορία των αγαθών, ε, των εμπορευμάτων. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, έχουμε να επενδύσουμε για όλα αυτά τα ωραία που ακούμε, τις τεχνολογίες. Πολλά κράτη-μέλη είναι χρεωμένα, υπερχρεωμένα ή στο χείλος της χρεοκοπίας. Επίσης αναφέρεται τις ε, ρυθμιστικές αρχές. Μπορεί πράγματι να είναι χρήσιμα, αλλά ξέρουμε στην καθημερινή ζωή πώς ε, λειτουργούν και πόσο επηρεάζονται από τις ομάδες πίεσης θα ήθελα να σχολιάσω αυτά που είπε ο Αυστριακός ε, συνάδελφος. Ε, ορισμένοι συνάδελφοί μου είπαν ότι το, το κόστος αυτών των προγραμμάτων είναι πάρα πολύ ψηλό. Η αγορά μπορεί να εκτιμάται σε 500 δις όμως, ορισμένα ψηφιακά προγράμματα μπορεί να συνδέονται ε, με τη διαφθορά και λόγω διαφθοράς που υπησέρχεται στα προγράμματα αυτά αυξάνεται το κόστος στο δεκαπλάσιο. Τι, τι θα κάνουμε επίσης με την ανακατανομή του εργατικού δυναμικού, με τις κοινωνικές επιπτώσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε τα πόδια μας στο έδαφος, να είμαστε πιο ορθολογικοί στη, στο σκεπτικό μας, πιο ρεαλιστές και να σκεφτόμαστε πάντοτε το κόστος. Μην... Υπάρχουν πάντοτε και αντίθετοι δείκτες σε αυτά που συζητάμε, αρνητικοί δηλαδή. Ε, ευχαριστώ. Πολλά ερωτήματα θέσατε και βέβαια πρέπει να απαντηθούν. Άρα ακόμα περισσότερη δουλειά μπροστά μας. Ο κύριος Ετσεβερία, Ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Ε, συγγνώμη που καθυστέρησα εδώ, αλλά είχα αλλού συναντήσεις ε, και με 14 στελέχη και πρόεδρους ε, των περιφερειών της χώρας μου. Είχα συναντηθεί πριν από λίγο για τις δυνατότητες αυτές του ηλεκτρονικού εμπορίου και τη σημασία για την Single Market Act. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε ότι πρόκειται για σημαντικό εργαλείο για θέσεις εργασίας καινούριου, για εμπιστοσύνη, για καλύτερο ανταγωνισμό, ανταγωνιστικότητα και εδώ θα μπορούσε να τονώσει το εμπόριο στην Ευρώπη. Η έξοδος από τη σημερινή κρίση έχει ψηφιακή μορφή κατά την απόψή μου και για συγκεκριμένο λόγο το λέω. Στην Κρακοβία είχαμε ζητήσει το φόρουμ για το Single Market Act και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή είμαστε παρόντες και το Συμβούλιο επίσης και ήταν ιδιαίτερα πλούσια η συζήτηση και είχα την δυνατότητα ακριβώς είχα την ευκαιρία να είμαι ο εισηγητής Τη ομάδα εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Να σα το πω σαφώς, η έξοδος από την κρίση έχει ψηφιακή μορφή γιατί προχωράμε σε μια ανευπροηγουμένων επανάσταση πέρα από την ε, βιομηχανική επανάσταση στο τέλος του 19ου αρχές 20ου αιώνα που έδωσε δυνατότητες στον 20ο αιώνα μετά. Τώρα ξεκινάμε πάλι πάνω σε αυτό και θα ήθελα να επωφεληθούμε από τη νέα αυτή επανάσταση. Έχει αλλάξει ακριβώς ε, ο τρόπος ε, συμπεριφοράς όλων των γενεών, ακόμα και εκείνες που είχαν γεννηθεί παλιότερα, έχουν γεννηθεί παλιότερα και το μέλλον περνάει από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στην Ευρώπη, όχι σε εθνικό επίπεδο, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, εντάξει, καλά τα πάει το ηλεκτρονικό εμπόριο, δεν αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα προβλήματα, όλο ένα και αυξάνεται αυτό, αλλά έχουμε προβλήματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί το συζητήσαμε σε αρκετές περιπτώσεις το θέμα αυτό. Εδώ υπάρχουν ε, εμπόδια ανάμεσα τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν μπορεί να εξαπλωθεί παντού σύμφωνα με το δυναμικό του χαρακτήρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και για το ίντερνετ και για το εκτό εμπόριο. Αναφερόμαστε σε ένα θέμα που αναπτύσσομαι και σαν να είναι το μέλλον ενώ δεν είναι πια μέλλον αλλού, είναι παρόν. Και θα ήθελα να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο συγκεκριμένο Είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη του πανευρωπαϊκού ηλεκτρονικού εμπορίου ή θα πρέπει να το αφήσουμε σκέτα σε εθνικό επίπεδο. Εδώ με απασχολεί αυτό. Μιλάμε πάντα για περισσότερη Ευρώπη, αλλά τι γίνεται. Δεν ξέρω. Μήπως θα έπρεπε να μιλάμε για λιγότερη Ευρώπη σε αυτό. νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να περάσουμε σε μια δεύτερη φάση και θα πρέπει να το συζητάμε βέβαια πάντως, αλλά τα ταυτόχρονα να ξεκινήσουμε ενέργειες για να ενισχύσουμε ακριβώς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το είπαμε με μια λέξη το σημαντικό θέμα είναι η εμπιστοσύνη. Χρειάζεται εμπιστοσύνη στο μέσον αυτό που δεν υπάρχει, ίσως δεν φαίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο επαρκώς στα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται και σύμφωνα με το δυναμικό του χαρακτήρα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να εργαστούμε ακριβώς και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ενισχύσουμε αυτό το εργαλείο στο οποίο πιστεύουμε και ολοκληρώνω την παρέμβασή μου κύριε Πρόεδρε για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε πια από την κρίση αυτή από την κρίση αυτή και η έξοδο από την κρίση έχει ψηφιακή μορφή επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά Ευχαριστώ που ήταν πραγματικά επί της ουσίας. Υπάρχει κάποιος που, άλλος που θέλει να μιλήσει παρακαλώ. Δεν υπάρχει άλλος που να θέλει να πάρει το λόγο, οπότε θέλω να ζητήσω από τον κύριο Μετζίντλο να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση η οποία θα έλεγα ήταν αισιόδοξη στην ανάλυση της ε, ψηφιακής, ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Υπάρχουν βέβαια ορισμένες πτυχές που ακούστηκαν αρνητικές και μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρανόησε ε, μερικά από αυτά τα οποία είπα. Όταν μιλάμε για 500 δις ε, ευρώ είναι το ποσό αυτό το οποίο θα ε, θα υπάρξει, θα δημιουργήσει όταν η ψηφιακή αγορά γίνει πραγματικότητα. Δηλαδή το 4% είναι το επιπλέον τα 507 δις από το συνολικό όγκο της ευρωπαϊκής αγοράς, της ενιαίας αγοράς. Και η Ευρωπαϊκή Κομισιόν έχει αναφέρει αυτήν τη δυνατότητα ανάπτυξης. Αναφέρθηκε βέβαια και το θέμα της διαφθοράς και δεδομένου ότι ασχολούμαστε εδώ με τις δημόσιες προμήθειες υπάρχει το στοιχείο, η δυνατότητα της διαφθοράς δεδομένου ότι όλες αυτές οι συμβάσεις γίνονται μεταξύ ανθρώπων. Ε, ε, βεβαίως υπάρχουν ρήτρες, υπάρχουν ε, πλαίσια προστασίας κατά της διαφθοράς αλλά είναι και η διαφθορά μία απειλή και μία πρόκληση, ειδικά όταν αναφερόμαστε στην υποδομή, στην εδραίωση της υποδομής. Ο Γάλλος συνάδελφος είπε ότι η Γαλλία είναι πρόθυμη να επενδύσει 25 δισεκατομμύρια στα, στις οπτικές ίνες. Και εμείς ε, οποίου εφαρμόζουμε πλέον ε, την ευρυζωνική πρόσβαση και τα ευρυζωνικά δίκτυα στην Πολωνία και μάλιστα έχει περάσει ένα ειδικό νομοσχέδιο που διευκολύνει την ε, παροχή ευρυζωνικών δικτύων. 1,5 δις ευρώ έχουμε επενδύσει ε, και είναι η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το πρόγραμμα. Αλλά Έχουμε άλλο, ψηφίστηκε άλλο ένα νομοσχέδιο που διέθεσε ένα επιπλέον δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι λοιπόν ε, ένα πρόγραμμα αυτό το οποίο ε, ήδη χρηματοδοτήθηκε, είναι στη φάση της υλοποίησης. Όταν μιλάμε για δημόσια χρηματοδότηση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν είναι τόσο εύκολο να δοθεί αυτή η χρηματοδότηση και να διοχετευτεί περιφερειακά και τοπικά. Πάρα πολλά πρέπει να γίνουν για να βελτιωθούν οι επενδύσεις στην ψηφιακή αγορά. Και πολλά μπορούν και πρέπει να γίνουν στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ελπίζω ότι θα ανταποκριθούμε στη μεγάλη αυτή πρόκληση. Υπάρχει και η νέα οδηγία για την ηλεκτρονική υπογραφή και πιστεύω ότι δεν θα αργήσει η υιοθέτησή της διότι αυτή η οδηγία είναι πάρα πολύ σημαντική. Στην Πολωνία πρόσφατα ε, είδαμε τις επιπτώσεις της οδηγίας αυτής, διότι πρέπει να τροποποιήσουμε το, τη δική μας νομοθεσία για την, εθνική, για την ψηφιακή υπογραφή ακολουθώντας ε, τις ε, διατάξεις της ε, οδηγίας αυτής η οποία ακόμα εκκρεμεί. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτή η οδηγία θα εφαρμοστεί, θα επικυρωθεί πολύ σύντομα διότι είναι πολύ σημαντική για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής και πολύ σημαντική για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Ευχαριστώ για τα συμπεράσματα της συζήτησης. Ευχαριστώ και όλους τους συμμετάσχοντες σε αυτήν την πολύ ε, χρήσιμη και ζωντανή συζήτηση και τώρα δίνω το λόγο στον πρόεδρο του ΙΜΚΟ, κύριο Χάρμπορ. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Εγώ θα προεδρεύσω κατά τη διάρκεια της τελευταίας ε, συζήτησης ε, σήμερα το πρωί για τις δημόσιες προμήθειες. Για, το, για τις δημόσιες προμήθειες είναι νερό το φυλάδιο. Επομένως, αν κάποια μέλη του, των Εθνικών Κοινοβουλίων θέλουν να πάρουν το λόγο, παρακαλώ συμπληρώστε το. Από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα ανακοινώσω και εγώ τα ονόματα, αλλά σίγουρα θα υπάρξει χρόνο και για άλλε παρεμβάσει. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ζήτημα για την ενιαία αγορά, την ιστορική αγορά, όχι μόνο για την δημιουργία μια αγορά, αλλά και επειδή η δημόσια προμήθεια είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, τομέας ε, για ε, την επίτευξη άλλων στόχων, όπω η πράσινη οικονομία, πιο δίκαιη οικονομία και πιο ανοιχτή οικονομία. Και αυτά αντικατοπτρίζονται και στην ικανοποίηση για την ε, τρέχουσα ε, ε τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Έχουμε δύο ε, εκθέσεις ε, ιδίας πρωτοβουλίας. Η συγκίτριά μας βεβαίως ε, είναι το κατάλληλο άτομο για να μας μιλήσει από αυτού. Υπάρχει το κείμενο, ε, το οποίο δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες αυτή τη στιγμή, αλλά σύντομα θα είναι στον ιστότοπο και θα μπορέσετε να το ε, κοιτάξετε. Θα καλέσω λοιπόν τη Heidi Ruler να ανοίξει ε, τη συζήτηση. Έχει το λόγο για πέντε λεπτά. Μετά έχουμε τον κύριο Γιωχάνσον από τη Σουηδία και την κυρία Φεσάιτσε από τη Λιθουανία. Και μετά Άντβες Φάβε από το ΕΛΚ. Δίνω λοιπόν το λόγο για πέντε λεπτά στην Χάντι Ρούλα. Ευχαριστώ. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Δημοσίων Προμηθειών χρειάζεται να επιδείξει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και διαφάνεια. Όμως σε αυτή την νομοθεσία ε, για τις δημόσιες προμήθειες υπάρχουν πολλά αμφιλεγόμενα και αντιμαχόμενα θέματα τα οποία δημιουργούν ε, μείωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και πολλές τριβές στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό ακριβώς ενσωματώθηκε στη στρατηγική του 2020. Είμαστε ικανοποιημένοι με την πράσινη βίβλο της Κομισιόν και τη διαδικασία αναθεώρησης. Καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι αυτή η αναθεώρηση πρέπει να γίνει μαλακά μαλακά. Αυτό το συζητήσαμε στην Κρακοβία την περασμένη εβδομάδα. Δεν χρειάζονται ξαφνικές ε, ενέργειες, αλλά μια απαλή, μια ήπια αντιμετώπιση της ε, αναθεώρησης αυτής. Η οδηγία θα πρέπει να σεβαστεί τις υπάρχουσες βασικές διατάξεις ε, τις διάφορες κατηγορίες, τις υπηρεσίες Α και Β, υπεργολαβίες κλπ. Όμως πρέπει να δείξει σαφώς ότι το νομικό πλαίσιο είναι εδρεωμένο και, ε, ε, και, και πιο διαφανές και ευέλικτο. Δεύτερον, καινοτομίες και αηφόρο εργασία, αιφόρος ανάπτυξη της αγοράς εργασίας, εκεί διαπιστώνουμε ότι για την καινοτομία και την αγορά εργασίας τα περισσότερα προσκόμματα βρίσκονται στους κανονισμούς, στις, ε, συγγνώμη, οδηγίες. Έχουμε αυτή τη στιγμή μία αντίφαση μεταξύ του φθηνό, της φθηνότερης προσφοράς και της καλύτερης προσφοράς. Ενώ αυτή τη στιγμή διαπιστώνει το Κοινοβούλιο ότι αυτή τη στιγμή προτιμάται η βέλτιστη προσφορά και όχι φθηνότερη προσφορά, η οποία χρησιμοποιείται μόνο σε ορισμένα προϊόντα. Αυτό είναι μια σωστή προσέγγιση. Θέλουμε να διευκολύνουμε ακόμα περισσότερο την ε, έγκριση των καλύτερων ε, προσφορών και χρειαζόμαστε περισσότερα πρότυπα για τη ρύθμιση αυτού του θέματος, αυτού του πλαισίου. Επίσης, δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο το προϊόν αυτό αυτό, αλλά και διαδικασία παραγωγής κατασκευής. Δηλαδή, τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, τεχνική ορολογία. Όλα αυτά σε μία αναθεώρηση πρέπει να ε, οριστούν σαφώς. Στις δημόσιες προμήθειες πρέπει να ε, υιοθετηθούν περισσότερα πρότυπα πρότυπα τα οποία είναι ανοιχτά, δηλαδή διευκολύνουν την πρόσβαση και επίσης η δημιουργία μας ε, ε, τράπεζες δεδομένων η οποία περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες ταυτοποίησης. Ε, το τρίτο, τρίτο στόχος είναι ένα σαφές πλαίσιο εποπτείας της αγοράς διότι σε πολλές διατάξεις είναι σαφές η εφαρμογή τους δεν είναι σαφή, δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα εφαρμοστούν. Θέλουμε μία καλύτερη χρησιμοποίηση και εφαρμογή της διαδικασίας διαβούλευσης, της διαδικασίας δημοσιοποίησης και την ε, αύξηση των κριτηρίων ε, στη διαδικασία δημοσίευσης και δημοσιοποίησης, διότι μέχρι τώρα ε, δεν έφταναν τα κριτήρια αυτά για την επιβολή της διαφάνειας. Θέλουμε επίσης να επιτρέπονται παράπλευρες προσφορές σε ένα μειοδοτικό διαγωνισμό, και τι δυνατότητα διόρθωσης λαθών. Βεβαίως, η διόρθωση των λαθών πρέπει να γίνεται βάσει καθαρών, σαφέστατων κριτηρίων διαφάνειας. Προτείνουμε η Κομισιόν να εξετάσει όλα τα κατόφλια τα οποία αξιών τα οποία προσφέρει, τα οποία προτείνει και να αυξηθούν οι τιμές, να αυξηθούν οι τιμές κατοφλίου. Δίδουμε περισσότερη σημασία στην πρακτική πλευρά, περισσότερη ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας, περισσότερη αξιολόγηση καθιερωμένων συστημάτων και μεθόδων, αυστηρότερη εποπτεία και έλεγχος, περισσότερη χρησιμοποίηση των υπαρχουσών δικτύων, των υπαρχόντων δικτύων και περισσότερη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος συναλλαγών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την εφαρμογή της αρχής Only Once, μια φορά μόνο, έτσι ώστε μόνο μια φορά να υποβάλουν όλη αυτή την τεκμηρίωση μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μην πνιγούν σε όλο αυτή το χαρτοβασίλειο. Προτιμούμε βεβαίως και θα το τονίσουμε μια ηλεκτρονική διαδικασία που θα διευκολύνει ακόμα περισσότερο και τους μικρομεσαίους και θα αποφύγουν τη γραφειοκρατία Πρέπει επίσης να εφαρμοστεί η αρχή ε, explain and apply, ε, εξήγηση και εφαρμογή και τέλος ηλεκτρονικές προμήθειες, ηλεκτρονικές αναθέσεις. Το σύστημα αυτό το ηλεκτρονικό θα πρέπει να σωματωθεί στις διατάξεις της ε, οδηγίας ε, μέχρι 15% δεν έχουμε ακόμα επιτύχει τους στόχους μας 15% των αναθέσεων γίνεται ηλεκτρονικά μόνο και θέλουμε οπωσδήποτε να αυξηθεί αυτό για να αυξηθεί η ηλεκτρονική ανάθεση πρέπει να λυθεί το θέμα της ηλεκτρονικής υπογραφής άρα πρέπει να περάσει η οδηγία αυτή το σοντιμότερο Πρέπει επίσης να είναι συμβατές οι διάφορες πλατφόρμες και διαλειτουργικές, διαλειτουργικότητα λοιπόν των ηλεκτρονικών πλατφορμών να βελτιωθεί και για να ε, ενισχύσουμε όλη αυτή την ηλεκτρονική πτυχή. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Heidi. που ανέφερες, ανέφερες μερικά από τις πιο σημαντικές πτυχές ενός ιδιαίτερα περίπλοκου ζητήματος. Καλό θα ήταν βέβαια να έχουμε και την ίδια την έκθεση. Πρέπει να βρούμε τρόπους να αυξήσουμε την δράση μας ε, στον τομέα των δημόσιων προμηθειών. Ας προχωρήσουμε τώρα στη συζήτηση. Καλό τον κύριο Γιωχάνσον από το Σουηδικό Κοινοβούλιο να πάρει το λόγο για τρία λεπτά. Κύριε Γιωχάνσον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Οι δημόσιες προμήθειες αποτελούν ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς και της κατανάλωσης. Ε, δίνουν ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα και στους καταναλωτές για τις περιβαλλοντικές τους επιλογές ε, και πολλούς άλλους τομείς. Είναι σημαντικό και εμείς να ε, εφαρμόζουμε τις αρχές της αναλογικότητας, της, των μη διακρίσεων, της διαφάνειας. στη Σουηδία στα προϊόντα, διατροφικά προϊόντα μόνο το 50% παράγονται στη χώρα μας. Γι' αυτό ε, στρεφόμαστε προς άλλες χώρες, όπως η Γερμανία κυρίως. Ε, και βεβαίως τους ευγνωμονούμε τους Γερμανούς αγρότες που παράγουν τα προϊόντα για εμάς. Ε, η Σουηδία έχει πληθυσμό 9 εκατομμυρίων ανθρώπων. Στον δημόσιο τομέα 3 εκατομμύρια γεύματα σερβίρονται κάθε μέρα ε, στα σχολεία, στους ηλικιωμένους, στα νοσοκομεία και ούτω καθεξής το επίπεδο της αυτοεξυπηρέτησης είναι πολύ χαμηλό ε, ή ακόμα και σε αυτές τις ε, περιοχές. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα για να το βελτιώσουμε, αλλά δεν έχουμε καταφέρει πολλά. Ε, για τις προδιαγραφές των προϊόντων είναι από τις πιο αυστηρές όλη την Ευρώπη. Για το κρέας, για παράδειγμα, έχουμε πολύ αυστηρές προδιαγραφές ε, για τα ζώα, τον τρόπο σφαγή τους και τον τρόπο που έζησαν πριν από αυτό. Ε, Βεβαίω, όταν υπάρχει παραβίαση των ε, ε, νόμων υπάρχουν κυρώσει, αλλά οι ίδιε αυτέ αρχέ αγοράζουν τρόφιμα από, ε, από εκτροφεί που, ε, διατηρούν τα ζώα του σε πολύ χειρότερε συνθήκε από αυτέ που έχουμε στη, στην Σουηδία. Είναι σημαντικό λοιπόν οι νόμοι να ε, διατυπώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουμε το ε, υψηλότερο επίπεδο προστασία του καταναλωτή, ε, ξεκάθαρε συσκευασίε για να ξέρουμε κι εμεί ε, τι ακριβώ αγοράζουμε. Ε, οι διατάξεις για την ευημερία των ζώων δεν είναι εναρμονισμένες αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, στις δημόσιες προμήθειες είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου το άρθρο 13 της ε, ε συνθήκης ε, όπου προβλέπεται ότι πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη η ευημερία των, και η υγεία των ε, ζώων. Οι εθνικέ νομοθεσίε δεν είναι πάντα ε, ξεκάθαρε και αυτό είναι δικό μα καθήκον να αυξήσουμε τη διαφάνεια. Πρέπει να νορμονίσουμε την προστασία των ζώων σε όλη την Ευρώπη, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των διακρίσεων που υπάρχει στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρονται αυτά τα στοιχεία και βεβαίως η ευζοία των ζώων και τα πρότυπα της ευζοίας των ζώων δεν είναι ευθύνη αυτή της επιτροπής αλλά υπάρχουν προτάσεις εναρμόνισης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Βερσάιτε από τη Λιθουανία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Ρίλε, για την έκθεσή της με το πολύ σημαντικό αυτό θέμα των δημοσίων προμηθειών. Τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι διαμέσου των προμηθειών αυτών ο κόσμος χάνει περίπου 400 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω διαφθοράς και πιστεύω ότι η διαφάνεια και η μάχη κατά της διαφθοράς είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Οι δημόσιες προμήθειες και ε, το σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών είναι ε, πάρα μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Ένα άλλο πρόβλημα που αναφέρεται στην γνωμοδότηση είναι η χαμηλότερη τιμή ε, σε, έναν ε, ε, δημόσιο, σε μια δημόσια προκήρυξη οι προσφορές με τη χαμηλότερη τιμή που πολλές φορές επιλέγονται. Εάν δούμε τον κατασκευαστικό τομέα και τη μακροπρόθεσμη προοπτική, διαπιστώνουμε ότι η, η, η παροχή των συμβάσεων, η ανάθεση των συμβάσεων στον μειοδότη δεν Οφέλησε πολλές φορές το έργο. Δεν είχε θετικά αποτελέσματα. Επίσης, απλουστευμένες διαδικασίες, προηγμένες τεχνολογίες και αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη όπως και οι μικρομισές επιχειρήσεις και η πρόσβασή τους στη, στους, στις προκηρύξεις αυτές. Η πρώτη τάσεις που περιλαμβάνει αυτή η έκθεση δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα των μικρομεσαίων. Δεν πρέπει να ανακαλύψουμε εκ νέου τον τροχό. Έχουμε θαυμάσια παραδείγματα διεθνώς, παραδείγματο χάρη από τις Ηνωμένε Πολιτείες που έχουν ένα πολύ ικανοποιητικό δίκτυο συμμετοχής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται και αναφέρονται στην αρχική σύμβαση. Γιατί λοιπόν δεν μπορούμε και αυτό να το υιοθετήσουμε. Χρειάζεται συγκεκριμένη δράση. Εάν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και να ενεργήσουμε ορθολογικά στη διαχείριση των ε, χρημάτων των φορολογούμενων, σε εθνικό επίπεδο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι κυβερνήσεις πολλές φορές είναι και οι μεγαλύτεροι εργοδότες. Άρα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτές τις πτυχές που ανέφερα, να τις μελετήσουμε για να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες και τους μακροπρόθεσμους στόχους και αποτελέσματα Επίσης πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα χρήματα των φορολογούμενων θα προσδώσουν τη θέμενη αξία. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κ. Σβάμπ. Του ΕΛΚ. Ο κ. Βαλκούνατς από τη Λιθανία και ο κ. Μπόνατς από το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Κύριο Σβάμπ, ευχαριστώ πρόεδρε η ευκαιρία αυτή να συζητήσουμε αυτά τα σημαντικά θέματα με τους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Τα θέματα της ενιαίας αγοράς. Η κυρία Ρίλη ανέφερε τα πιο σημαντικά σημεία της έκθεσης και γι' αυτό θα αναφερθώ ε, σε θέματα τα άλλα που μας απασχολούν και που άπτονται του του πλαισίου δημοσίων προμηθειών και θα αναφερθώ σε κάτι που είπε ο Λιθουανός συνάδελφος. Τα χρήματα των φορολογούμενων. Θα πρέπει τα χρήματα των φορολογούμενων να, δείξουν, να χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να αποδώσουν ένα δημόσιο όφελος στο πλαίσιο αυτό των δημοσίων προμηθειών. Γι' αυτό και οι προσφορές όλες αυτές και οι προκηρύξεις πρέπει να είναι σωστές και διαφανείς θα ήθελα λοιπόν να πω στους συναδέλφους ότι υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα για τη βελτίωση της υποδομής, της, κοινωνίας, της κοινωνίας, του, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε οι δημόσιες προκηρύξεις να προκηρύσσονται σωστά από αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τη λήψη των αποφάσεων, από τους αρμόδιους δηλαδή και όχι από άσχετους οι οποίοι εμπλέκονται και εφαρμόζουν άλλα κριτήρια τα οποία δεν έχουν σχέση με την ουσία των ε, διαγωνισμών των προμηθειών αυτών. Διότι, ε, όπως είπε στο τέλος, τα χρήματα των φορολογούμενων πρέπει να, προσφέρουν θέμενη αξία. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το θέμα δεν έχει προβληθεί όσο θα έπρεπε, διότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο χρήσης των, ε, ε, των χρημάτων των φορολογούμενων. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την, τα επιχειρήματα της Κομισιόν η οποία τονίζει πάντοτε τα ωφέλη της ενιαίας αγοράς. Άρα λοιπόν αυτό το πλαίσιο των φορολογούμενων και των χρημάτων τους και πώς διατίθενται δεν έχει φωτιστεί αρκετά. Πρέπει να χρησιμοποιούμε περισσότερο τη μέθοδο της κλήρωσης έτσι ώστε να μπορούμε να δώσουμε καλύτερες ευκαιρίες στις μικρομεσαίες να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Κλήρωση λοιπόν, να χρησιμοποιηθεί καλύτερα. Δεύτερον, συζήτησα με έναν συνάδελφό μου, ο οποίος στην περιοχή του γίνεται ένα, μια προσφορά για ένα νοσοκομείο ε, και πήραν πολλές προσφορές ε, στις προκηρύξεις από την περιοχή του της Βασιλείας αλλά από καμία άλλη χώρα. Ε, ε, θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω γιατί δεν έχουμε μια ευρύτερη υπερσυνοριακή συμμετοχή στις δημόσιες προκηρύξεις. Ε, δυστυχώς αυτό δείχνει ότι η ενιαία αγορά δεν λειτουργεί ακόμα σωστά όπως τα θέλαμε. Άρα λοιπόν πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε, σε λύσεις, σε προτάσεις λύσεων και να ξεπεράσουμε τα προσκόμματα σε αυτή την ενιαία αγορά πρέπει να, ε, ε, ε, αυτή η αγορά πρέπει να είναι ανοιχτή έτσι ώστε να μπορούν και διασυνοριακά να συμμετάσχουν ενδιαφερόμενοι στις δημόσιες προμήθειες και όχι μόνο σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βαλκούνας στην Τελφάνεια. Uh, Έχετε τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έγινε αναφορά στην πράσινη βίβλο. Ελπίζω να μην πρόκειται για την πράσινη βίβλο του Καντάφη, του πρώην ηγέτη της Λιβύης. Επίσης, οι διατάξεις ε, που συζητούμε να εφαρμοστούν στην πράξη. Αυτό θα ωφελήσει τους ε, πολίτες μας. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δημιουργήσουμε, μάλλον να αναθρέψουμε ε, συνειδητοποιημένους και ε, ε έντιμους πολίτες που δεν θα θέλουν να κλέψουν. Διαφωνώ λοιπόν με τον ε, συνάδελφο από τη Λιθουανία. ότι πρέπει να καταργήσουμε τις χαμηλότερες τιμές. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και άλλα κριτήρια. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αναλύσουμε το ε, ιστορικό το αρχείο που έχουμε από, τους, από τις, ε, τις προσφορές της εταιρείε, να εξετάσουμε τα, τα βιβλία των εταιριών, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτές τις επιχειρήσεις, να ε, καταρτήσουμε ένα κατάλογο κριτηρίων. Και νομίζω ότι οι επιθεώρηση εργασία σε όλες τις ε, χώρες μπορούν να αναλάβουν αυτό το καθήκον. Μπορούμε επίσης να αξιοποιήσουμε την την φορολογική αστυνομία. Ε, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή ε, βάση δεδομένων όπου μπορούμε να βρούμε ε, πληροφορίες για, τα, για, τα, για όλες τις επιχειρήσεις. Να υπάρχει ένα αρχείο δηλαδή για όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Για να δούμε αν πρόκειται για αξιόπιστες ή μη επιχειρήσεις. Και τέλος, χρειαζόμαστε τα ονόματα αυτών των επιχειρήσεων για να ξέρουμε ποιες από αυτές ε, είναι αξιόπιστες. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Βαλκούνας. Επόμενος είναι ο κύριος Βανατσίν από το Ιταλικό ε, Κοινοβούλιο, μετά η κυρία Βάιλερ από τους Σοσιαλδημοκράτες, και μετά η κυρία Γκομάς από τη Γαλλία. Ευχαριστώ. <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε αυτό το θέμα της εσωτερικής αγοράς, η ε, διαγωνισμό του δημοσίου είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Όλοι πιστεύουν στην Ευρώπη ότι θα βγούμε από την κρίση, όπως το είπε και ο κύριος Ρισέ σήμερα το πρωί που είναι διαρθρωτική. Άρα λοιπόν χρειάζονται πολλές και διάφορες παρεμβάσεις. Όλα αυτά θα επιτευχθούν πρώτα απ' όλα με την οργάνωση μιας κατάλληλης υποδομής και με νέα δημόσια έργα. Και έτσι από φαινός φαίνεται κάτι το ιδιαίτερα εύκολο, αλλά δημιουργεί και προβλήματα και διαβάσαμε με ιδιαίτερη προσοχή την πράσινη βίβλο της Επιτροπής. Ε, κυβέρνηση πρώτα απ' όλα και μετά στις αρμόδιες επιτροπές ε, του Κοινοβουλίου και της ε, Γερουσίας. Το εξετάσαμε στο αρμόδιο τμήμα, οργανώσαμε ακροάσεις, συναντήσεις πολλές για το θέμα αυτό και μπορούμε να σας πούμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να συντάξουμε μια γνωμοδότηση όπως επίσης να υποβάλουμε και διάφορες προτάσεις για την πράσινη αυτή βίβλο που ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θεωρούμε. Ένας διαγωνισμός του δημοσίου φαίνεται, μια προκήρυξη του δημοσίου φαίνεται ότι θα πρέπει να ανταποκρίνεται και ανταποκρίνεται σε περισσότερο οικολογικές ανάγκες. Πρώτα απ' όλα τα χαρακτηριστικά αυτού του διαγωνισμού θα πρέπει να είναι η διαφάνεια, η ταχύτητα αυτής της προκήρυξης και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε αναταραχές από όσους θέλουν μέσω διαφθοράς να κερδίσουν αυτούς τους διαγωνισμούς και να μπει στη μέση και το οργανωμένο έγκλημα που δυστυχώς τώρα πια είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα να πω και παγκόσμιο θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρξουν και μέσα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που σε αυτές τους διαγωνισμούς θα ήθελαν να συμμετάσχουν και που ενώ έχουν τη διάθεση δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό λοιπόν. Εδώ στην Ιταλία 2008-2009 στο ξεκίνημα της θητείας ε, συντάξαμε ένα κώδικα για αυτό τους διαγωνισμούς που είναι ένα ευέλικτο εργαλείο και που προκάλεσε μια αλλαγή όσον αφορά τους διαγωνισμούς στην Ιταλία. Και γι' αυτό ακριβώς και το εργαλείο αυτό το γνωρίζουν όλοι νομίζω το project financing αυτό το σχέδιο το οικονομικό, δημοσιονομικό και δύσκολο όμως είναι οποιαδήποτε χώρα, να έχει τα χρήματα ακριβώ για να χρηματοδοτήσει ένα δημοσιοέργο. Πολλοί ιδιώτες θα ήθελα να συμμετάσχουν πια. Και εδώ έχουμε αυτό το project financing τρίτης γενιάς και έχουμε τη δυνατότητα τώρα να βάλουν κεφάλαια ιδιώτες για να παρεύουν, να συμμετάσχουν, να δημιουργήσουν την υποδομή και σιγά σιγά να μπουν και στο κεφάλαιο αυτό, μάλλον να ε, πάρουν πίσω τα κεφάλαιά τους μέσω της διαχείρισης. Θα πρέπει να το ξυπήσουμε αυτό το μέσο και εργαλείο έτσι να μπορέσουν να βρουν τα κράτη, τα κονδύλια, τα κεφάλαια που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να διαθέσουν από μόνα τους. Σας ευχαριστώ. Μικρόφωνο παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ και σήξατε και πάλι ένα πολύ σημαντικό θέμα την οικονομική και κοινωνική πλευρά των δημοσίων προμηθειών. Κυρία Βάιλερ από τους Σοσιαλδημοκράτες. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προλαλήσαντες, συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είναι μια πολύ σημαντική βάση αυτή η συζήτηση για μας και θα ήθελα να προσθέσω κάτι γενικά για την σημερινή κατάσταση. Η Κομισιόν θα παρουσιάσει μια πρόταση οδηγίας το Δεκέμβριο επί τη βάση της έκθεσης Ρούλε, την οποία έχουμε υπερψηφίσει και αυτό, αυτό είναι σίγουρο ε, αυτό το γεγονός και θα κοιτάξουμε τις προτάσεις της Κομισιόν από κοντά το Δεκέμβριο. 18%, 17-18% του ΑΕΠ είναι δημόσιες προκηρύξεις, δημόσιες προμήθειες, οφείλεται στις δημόσιες προμήθειες και αυτό το υψηλό ποσοστό καταδεικνύει ότι θα πρέπει να γίνουν από πλευρά κρατών μελών πολλά προγράμματα, θα γίνουν ακόμα πολλά προγράμματα επενδύσεων, άρα αυτό το ποσοστό 17% θα αυξηθεί ενδεχομένως. Ευχαριστούμε την κυρία Ρούλε για την δουλειά που έκανε μέχρι τώρα για το σχέδιο έκθεσης και την ευχαριστούμε για τις προτάσεις της, για την ευρύτερη συμμετοχή των μικρομεσαίων. Ε, είναι γεγονός ότι στα κράτη-μέλη οι μικρομεσαίοι είναι η κινητήρια δύναμη. Όχι τόσο οι μεγάλες και τρανές επιχειρήσεις, γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να τους επιτρέπουμε και να τους διευκολύνουμε τη συμμετοχή το δεύτερο σημείο το οποίο σίγουρα σας απασχολεί και σας από την εμπειρία σας είναι η συμμετοχή των διασυνοριακών σε, σε διασυνοριακά προγράμματα, διασυνοριακά έργα. Ασφαλώς εδώ μιλάμε για περιφέρειες που βρίσκονται κοντά στα σύνορα κρατών μελών. Τώρα κάτω από το 2% είναι η συμμετοχή, η διασυνοριακή στις ε, προκηρύξεις για δημόσιες προμήθειες. Δεν είναι τόσο το γλωσσικό πρόβλημα, διότι οι περισσότεροι μπορούν να συνεννοηθούν στα αγγλικά. Γιατί λοιπόν, ποια είναι ακριβώς τα προσκόμματα. Τώρα ο πρόεδρος είπε, αναφέρθηκε ήδη στην, σε προκηρύξεις και αναθέσεις με κριτήρια πράσινα. Εντάξει, αυτό γίνεται εδώ και χρόνια. Αυτό όμως που λείπει είναι η εφαρμογή των κοινωνικών κριτηρίων σε περιπτώσεις όπου η αγορά εργασίας λειτουργεί δυσμενώς, όπου υπάρχουν κατάσπαρτα κοινωνικά κριτήρια, πρέπει όλα αυτά να τα συγκεράσουμε. Αυτό το κατάλαβε η Κομισιόν στη στρατηγική 2020. Χρειαζόμαστε στις δημόσιες προκηρύξεις να παρουσιάζονται κίνητα, να παρουσιάζονται ε, γιατί, γιατί, να ανατηρούνται και να γίνονται σεβαστές οι διατάξεις για το στοιχείο του φύλου, τη συμπερίληψη της διάστασης του φύλου, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας Θέλουμε επίσης την τοπική διάσταση ε, να λαμβάνεται υπόψη, δηλαδή οι συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης που λαμβάνουν τις αποφάσεις και το μυαλό έχουν και την δυνατότητα κρίσης αλλά μπορούμε την κινητήρια δύναμη να την αναθέσουμε στην Κομισιόν. Αυτό μπορούμε να το, να το αφήσουμε στα χέρια της Κομισιόν. Πώς θα μπορέσει να πλουστεύσει τις διαδικασίες, να κάνει οικονομία στη χρησιμοποίηση των πόρων και ορθολογική χρήση. Αυτές τις βασικές γραμμές λοιπόν μπορούμε να τις, να τις μελετήσουμε από τις προτάσεις της Κομισιόν για να σηματοθούν στη νέα νομοθεσία. Σας ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ. Κύριε Παπαγεωργίου και μετά ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσω σε αυτά που είπε κύριε Βάιλερτ για πώς θα συμμετάσχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να απαντήσω το εξής. Οι δυσκολίες τους ε, είναι το περίπλοκο αυτών των προκήρυξεων και ίσως ε, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία το πώς κανείς μπορεί να ανταποκρίνεται όπως πρέπει σε αυτό και να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τουλάχιστον να συμμετέχουν, ε, να κερδίζουν χρόνο, να απλοποιείται το έργο τους. Άρα λοιπόν αυτή η διαδικασία μιας πιστοποίησης ώστε να απλουστευτούν οι διοικητικές διαδικασίες μέσω αυτής της στο Μοζέλα μεταξύ Λουξεμβούργου και Γερμανίας έχουμε δυσκολίες εκεί. Εκεί είναι η γλώσσα η δυσκολία γιατί γίνονται οι αυτές στα γερμανικά και οι δικές μας μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Λοιπόν και από γλωσσικής πλευράς διευκολύνουμε την κατάσταση και τις συνθήκες για την ιδιαίτερα περίπλοκη για τις μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις. Και επίση η γαλλική θέση ποια είναι για τις υπηρεσίες που προσφέρονται και βασιζόμενοι στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει αυτό είναι βάση της συνθήκης ίση αντιμετώπιση των υποψηφίων και διαφάνεια. Για να δούμε τώρα μια διαφάνεια επαρκής για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν η μια την άλλη. Η διαδικασία, η υποψηφιότητα όλων εκείνων πραγματικά ενδιαφέρονται με συγκεκριμένα πράγματα. Όλα αυτά που τα γνωρίζουν ακριβώς οι ενδιαφερόμενοι. Ίσως ε, μια ρύθμιση ακριβώς θα άνοιγε ακόμα περισσότερο το θέμα της διαχείρισης ε, στην αγορά, στον ανταγωνισμό και οι στόχοι της ιστορικής αγοράς ώστε ο καθένας να μπορέσει να προσφέρει υπηρεσίες ποιοτικές, χαμηλές λογικές όμως τιμές, με ίσο ανταγωνισμό, δίκαιο ανταγωνισμό, φαίνεται ότι θα μπορούσε, μπορεί να έχει επιτευχθεί και αρκετοί ήδη καλύπτονται από τις ειδικέ ευρωπαϊκές ρυθμίσεις, είτε με άλλους τομείς, αλλά είτε φορείς ούτε άλλος ζητάει άλλη περαιτέρω ρύθμιση. Αυτό το είχε τονίσει η έκθεση για την εσωτερική αγορά και την προστασία καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 10 Μαΐου του 2010 για το τι γίνεται με τις εσωτερικές αγορές και λέγεται ότι πρόταση νομοθετικού χαρακτήρα σχετικά με αυτή τι υπηρεσίες θα μπορούσε να γίνει για να αποφευχθούν στρεβλώσει τη εσωτερική αγοράς και τονίζεται ότι καμία στρέβλωση δεν ε, διαπιστώθηκε μέχρι τώρα και νομοθετική πράξη σχετικά με αυτές τι υπηρεσίες προσφέρονται δεν θα ωφελούσε από τη στιγμή που δεν θα αποσκοπούσε σε μια σαφή βελτίωση τη λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Γι' αυτό ακριβώ η γαλλική κυβέρνηση ε, ε, ανέλαβε νομίζω ε, θεωρεί ότι όλα αυτά που ισχύουν τώρα είναι τα κατάλληλα και ισχύουν ακριβώς μέσω του κοινοτικού δικαίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτό που είπατε. Ε, γιατί έρχεται πιο κοντά και στην γνωμοδότηση αυτή. Εμείς βέβαια αναμένουμε απάντηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Παπαγεωργίου για τρία λεπτά, μετά ο κύριος Κότσμαν και μετά ο κύριος Μιλέρ. Κύριε Παπαγεωργίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο πιο ασφαλής τρόπος για να αποφύγουμε αδικήματα, αδιαφάνειες και απάτες στις ε, δημόσιες προμήθειες είναι η συστηματική και εκτεταμένη δημοσιοποίηση και δημοσίευση των διαγωνισμών, αλλά πιστεύω και των αποτελεσμάτων αυτών των διαγωνισμών. Και φυσικά με χρήση του ε, διαδικτύου και της ηλεκτρονικής, όπως αν είναι και ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Όμως πάντα υπάρχει μια πτυχή, ωραία, η συγκίτριά μας μας είπε ότι θα πρέπει να υπάρχουν πρότυπα, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στο διαγωνισμό, αλλά συνήθως ο διάβολος κρύβεται στις παραλαβές αυτών των προϊόντων. Πολλές από τις συναλλαγές έχει παρατηρηθεί ιστορικά ότι γίνονται στις παραλαβές των προϊόντων και εκεί ο έλεγχος είναι πλημελής ή των υπηρεσιών. Ε, που καλούνται να αποκαλείται να αγοράσει ένα δημόσιο. Άρα θεωρώ ότι εκεί που να υπάρχει μια μεγάλη πρόβληψη επίσης στην ελεκτική διαδικασία και της παραλαβής των προϊόντων και ε, του ελέγχου για την ποιότητα, αν τηρούν τα στάνταρς, αν είναι στο, στα όρια των προτύπων. Θέλω επίσης να ε, σχολιάσω λίγο το πρόβλημα των μικρομεσαίων. Είναι δεδομένο ότι δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις δημόσιες προμήθειες. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, επειδή ο όγκος των ε, προμηθειών είναι μεγάλος, επειδή οι διαγωνισμοί είναι μεγάλου ύψους διαγωνισμοί, ε, προσκρούν στην ε, μία έκδοση εγγυητικών και ζητούνται εγγυητικές τραπεζών. Συνήθως οι τράπεζες σε μικρές επιχειρήσεις, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν εκδίδουν εγγυητικές. Είναι ένα από τα τεσσαβαντάζ και ένα, και ένα σημείο δυσκολιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ίσως εκεί πρέπει να προστρέξουμε σε πάγιες ε, λειτουργίες όπως πρόβλεψη για κοινοπραξίες, συμπράξεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή σπασίματος των διαγωνισμών κατά την τμηματική παράδοση και παραλαβή των υπηρεσιών των προϊόντων. Είναι δύο, ε, για παράδειγμα, πρόχειρες σκέψεις που κάνω για το πώς μπορούν να διευκολυθούν. Διότι όταν κάνεις μια μεγάλη προμήθεια σε ένα στρατό ή σε νοσοκομεία ο όγκος είναι μεγάλος, συνήθως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επαναλαμβάνω, δεν έχουν εγγυητικές επιστολές, δεν τις παρέχονται από τις τράπεζες και όταν ζητείτε να παραληφθούν ε, unblock, πάλι και εκεί δυσκολεύουν. Αν υπάρχουν όμως διαδικασίες κοινοπρακτικής λειτουργίας πολλών μικρομεσαίων ή πάντα με τις εγγύησεις των τραπεζών ή επαναλαμβάνω τμηματικής παράδοσης αυτών των προϊόντων με όλα τα άλλα που προείπαμε νομίζω ότι μπορεί να διευκολυθούν. Προφανώς και οι συνάδελφοι αλλά και όλοι εμείς και όσοι ιδιαίτερα είχαν εμπειρία από επιχειρήσεις και ιδιαίτερα συναλλαγές με δημόσιους οργανισμούς θα έχουν να προσθέσουν στην συνέχεια ή και σε άλλες διαδικασίες πολύ πιο περισσότερες ιδέες για τις μικρομεσαίες για να μην μείνει λόγος κενός και ναι μεν πρόθεση η διάθεσή μας να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες αλλά στην πράξη όπως λένε τις πράγματα που λένε οι δικηγόροι δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαγεωργίου και πιστεύω ότι συμφωνούμε απόλυτα για τις μικρομεσές και χαίρομαι που έχουμε την υποστήριξή σας σε αυτό το σημαντικό θέμα και το οποίο περιλαμβάνεται στις προτάσεις της κυρίας Ρίλε. Ο κύριος Κρόιτσμαν από την Άλντε. Τρία λεπτά. Ο κύριος Μίλε και ο κύριος Βέστλουντ μετά και η κυρία Κοράθα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Κρότσμαν, συνάδελφος. Ευχαριστώ, πρόεδρε, αξιότιμοι, αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι. Θέλω ξανά να ευχαριστήσω την Πολωνική Προεδρία που αναγνωρίζει τη σημασία μιας ε, αναπτυσσόμενης ενιαίας αγοράς και τη σημασία που έχει για την εξασφάλιση της ευημερίας και της αναζωγόνησης της Ευρώπης πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό της ενιαίας αγοράς ε, στο 100%. Θέλω λοιπόν για να γίνει αυτό να τονίσω τρεις τομείς. Απλούστευση των διαδικασιών και ελαστικότητα, την δημιουργία σωστών κριτηρίων για την ανάθεση και την ευρεία συμμετοχή και πρόσβαση στις προκηρύξεις. Η απλούστευση λοιπόν των κανονισμών διευκολύνει την εξέλιξη των διαβουλεύσεων, των διαπραγματεύσεων. Εγώ σας είπα ότι δεν έχω τίποτα εναντίον της απλούστευσης ε, και ε, των διαδικασιών των δημοσίων προμηθειών διότι όσο πιο περίπλοκες είναι οι διαδικασίες τόσο πιο εύκολο είναι να παρισφρήσει το στοιχείο της διαφθοράς. Ε, το είχαμε συζητήσει αυτό το 2007-2008 και όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό σε αυτό τον τομέα χρειάζονται κάποια χρονική περίοδο να προσαρμοστούν. Όμως αυτή η μεταβατική περίοδος πρέπει να εξασφαλίζει πρώτον διαφάνεια, δεύτερον αποφυγή διακρίσεων. Επίσης πρέπει να δημοσιεύονται ε, σαφέστατα τα αποτελέσματα των διαγωνισμών αυτών ώστε να ξέρουν και οι χαμένοι γιατί έχασαν. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται μία προκήρυξη διαγωνισμού μετά μία ανάθεση και εν συνεχεία να γίνονται ε, παράπονα και προσφυγές των άλλων συμμετασχόντων χωρίς να ξέρουν ακριβώς τους λόγους για τους οποίους ανατέθηκε στον ΑΒΓ και γιατί αυτοί χάσανε. Λοιπόν, διαφάνεια. Συνεχώς επανερχόμαστε στη διαφάνεια. Όσον αφορά τώρα την αύξηση των, ορο... αξιών κατοφλίων για τις ευρωπαϊκές προκηρύξεις, εδώ υπάρχουν υπέρ, γνώμες υπέρ και κατά. Ε, δεδομένου ότι δεν έχουμε τόσες πολλές προσφορές από τρίτα, τρίτους συμμετέχοντες, από διασυνοριακές προκηρύξεις δηλαδή, δεν βλέπω το λόγο γιατί να αυξηθούν αυτά τα όρια η Κομισιόν θα πρέπει να μας αποδείξει πρώτα ότι τα σημερινά όρια, τα σημερινά πλαφόν δεν είναι επαρκή πριν προτείνει μία αλλαγή των ορίων αυτών. Τρίτον, τα κοινωνικά κριτήρια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να συμπεριληφθούν κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά, αλλά σωστά, με το σωστό τρόπο. Υποστηρίζω την πρόταση της ε, κυρίας Ρούλε να ε, επιλέγονται πάντοτε τα, με κοινωνικά κριτήρια ε, οι, διαγωνισμοί. Δηλαδή να επιλέγεται ο, εκείνος ο οποίος έχει κάνει την πιο σωστή κοινωνική ε, πρόταση από κοινωνική πλευρά και να μην λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μειοδότες, οι χαμηλότερες τιμές επειδή έχει προχωρήσει η ώρα και επειδή πολλά ελέγχθησαν για τις μικρομεσές Συμφωνώ απόλυτα με την μεγαλύτερη συμμετοχή και πρόσβαση των μικρομεσαίων. Δεν είναι εύκολο αυτό. Η κυρία Βάιμπερ έκανε προτάσεις, άλλες ιδέες ακούστηκαν πολύ σωστά. Έχουν οι μεγάλες εταιρείες, όπως και να το κάνουμε, πλεονέκτημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, κύριε Κρότσμαν. Ο κύριος Μίλερ, από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, πολύ. Ο τομέας των δημόσιων ε, προμηθειών είναι ένα ευαίσθητος τομέας. Ε, σημαντικό ζήτημα το οποίο θίγουμε εδώ σήμερα. Υπάρχουν προβλήματα διαφθοράς, ε, απάτης και καχυποψίας βεβαίως και σε αυτό το θέμα. Βάσει βεβαίως των προσωπικών τους εμπειριών. Από την άλλη έχουμε και πολιτικές διαφωνίες στο ιστορικό επίπεδο για την ομοθεσία. Μετά μιλάμε για τα χρήματα των φορολογουμένων. Αν χαθεί η εμπιστοσύνη στην χρήση των ε, χρημάτων αυτών των φορολογουμένων, τότε υπάρχει πρόβλημα γιατί και οι ίδιοι οι πολιτικοί θα χάσουν την αξιοπιστία τους. Τι είναι μεγάλη μας ευθύνη λοιπόν. Ε, τα εθνικά κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία γι' αυτό και χρειαζόμαστε και βοήθεια. Ε, χρειαζόμαστε μια ενιαία αναρμονισμένη ε, νομοθεσία που θα μας βοηθά στην εφαρμογή των μέτρων αυτών. Για παράδειγμα, πώς μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Μία πτυχή που είναι πολύ σημαντική, πολλά κρατημέλη σίγουρα θα το έχουν βιώσει, ε, οι προσφορές στις δημόσιες προμήθειες ε, για την δημοσιοποίηση ε, και την ανακοίνωση της προσφοράς. Αυτό θα γίνεται με διαφανή τρόπο και να είμαστε σίγουροι ότι οι προσφορές γίνονται από εταιρείε με καθαρό μητρό γιατί υπάρχουν ε, βεβαίω ε, επιχειρήσει που κάνουν πολύ ενδιαφέρουσε ε, και ελκυστικέ προσφορέ, αλλά δεν ξέρει ποιο κρύβεται από πίσω. Τίποτα δεν ξέρει για αυτέ τι επιχειρήσει. Πρέπει λοιπόν να το, να το επιλύσουμε αυτό το θέμα. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τι απάτε. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι ε, έχουν καθαρό μητρό αυτέ οι επιχειρήσει. Δεύτερον, για τι μικρέ και μισέ επιχειρήσει. Συνήθω είναι να λαμβάνουν μια υπεργολαβία, αλλά τίποτα παραπάνω. Για μα είναι σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια και σε αυτό. Δημόσιες πληροφορίες. Για παράδειγμα, κάνει κάποιος μια προσφορά. Πρέπει να παρέχουν πληροφορίες. Με ποιους θέλουν να συνεργαστούν. Γιατί πολύ συχνά όταν έχουμε μεγάλα επενδυτικά προγράμματα, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χάνουν γιατί δεν έχουν τα, κατάλληλα, τους κατάλληλους πόρους και παράλληλα... Ε, πέφτουν θύματα απάτη. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια, γιατί αυτό θα βοηθήσει τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Κάτι άλλο το οποίο ήθελα να αναφέρω, μιλήσαμε για την επικουρικότητα και την ευθύνη των κρατών μελών. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε παραπέρα από αυτό. Το κόμμα μου είναι ε, οικολογικό. Έχουμε υποβάλει ψήφισμα στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο για ακριβώς αυτό το σημείο πριν την δημοσιοποίηση της, ε, του διαγωνισμού θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και της τοπικής κοινωνίας. Ε, τα ενδιαφερόμενα μέλη στην τοπική κοινότητα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Σε μια μικρή πόλη θέλουμε να κάνουμε ένα κατασκευαστικό έργο. Πρέπει να μιλήσουμε με την κοινωνία των πολιτών, του επαγγελματίε, τι επαγγελματικέ οργανώσει, να ζητήσουμε τι δικέ του απόψει πριν τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού. Ιδάλω χάνουμε και πάλι την εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτές τις πολύ πρακτικές προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία σας και ο κύριος Βέστλουντ από το Σουηδικό Κοινοβούλιο και, και εν συνεχεία eh, Ευχαριστώ λέει ο κύριος Βέστλουντ Μιλώντας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πιστεύω ότι η καλύτερη συμβουλή που μπορούμε να δώσουμε σε αυτή την Επιτροπή είναι να μειωθεί η γραφειοκρατία. Συνεχώς αυτό μας αναφέρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν ε, μιλάμε μαζί τους. Πάντοτε πρέπει λένε, μας λένε να, έχουμε ένα δικηγόρο, ένα νομικό σύμβολο δίπλα μας για να μπορέσει να μας εξηγήσει αυτές τις διαδικασίες των διαγωνισμών. Λοιπόν, κάντε τα πράγματα πιο εύκολα. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερο, το γεγονός ότι προτείνουμε να σπάσουν οι διαγωνισμοί αντί για έναν μεγάλο ε, 4-5 ή 2-3 μικρότερες προκήρυξεις. Αυτή μπορεί να είναι μια καλή ιδέα. Αλλά ο λόγος για τον οποίο ζήτησα να μιλήσω είναι επειδή είπε ο συνάδελφός μου, Γιώχανσον, ότι πρέπει να υιοθετήσουμε περισσότερα κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά πρέπει οπωσδήποτε να παρουσιάζουμε τα κριτήριά μας ξεκάθαρα. Δεν αρκεί να λέμε θέλουμε καλή προστασία των πολιτών, καλή προστασία του περιβάλλοντος, αλλά στη διαδικασία ε, δημοσίων διαγωνισμών δεν θα απαιτούμε την τήρηση αυτών των κριτηρίων. Αυτή δεν, η αντίφαση δεν είναι σωστή. Ένα άλλο στοιχείο που οπωσδήποτε πρέπει να συμπεριληφθεί στις δημόσιες προκηρύξεις είναι το κοινωνικό κριτήριο πρέπει να ε, συζητάμε. Όπως γίνεται και στις συλλογικές συμβάσεις και σε άλλες ε, συμφωνίες. Λαμβάνεται υπόψη το κοινωνικό κόστος, η κοινωνική διάσταση. Δεν θέλουμε να γίνεται μια διαδικασία ε, διαγωνισμού, δημοσίου διαγωνισμού που να ωφελεί μια συγκεκριμένη ομάδα στην κοινωνία. Έτσι θα δημιουργήσουμε διακρίσεις, θα, δημιουργηθεί, θα υπονομεύσουμε την αγορά εργασίας την, ε, τους μισθούς και τις αμοιβέ κλπ. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ξεκάθαρα κοινωνικά κριτήρια στα οποία να μπορούν να, να αναφέρονται οι προκυρήσοντες και οι διαγωνιζόμενοι. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο. Τι ζητάμε, πώς θέλουμε να γίνει αυτό το ζητούμενο και τι στόχους επιδιώκουμε. Ανοιχτή πρόσβαση και διαφάνεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος της ε, συζήτησης. Να αναφέρω τους τελευταίους ομιλητές. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτς θα λάβει το λόγο, μετά ο κύριος Φίστας. Μου δίνετε το λόγο. Ναι, μισό λεπτό. Είπα ότι θα διατρέξω εν συντομία τον κατάλογο των ομιλητών. Έκλεισε λοιπόν ο κατάλογος ομιλητών. Γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε μέχρι τις 12.30. Χουίς Τσάς, και τέλος κυρία Τούν. Αυτό είναι ο κατάλογο ομιλητών. Λυπάμαι που δεν έχουμε χρόνο για περισσότερους. Και η κυρία Μίλλερ θα συνοψίσει στο τέλο. Παρακαλώ, αυτό το λόγο. Ευχαριστώ δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνει ε, μια συζήτηση μεταξύ Σουηδών, αλλά με ενέπνευσε το σχόλιο του συναδέλφου ε, κ. Γιώχανσον και είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι δεν είμαστε υπέρ του διατροφικού ε, εθνικισμού. Δεν μπορείτε να κατηγορείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν η Σουηδία ή άλλο κράτος μέλος έχει διαφορετικές ερμηνείες ή, ή περαιτέρω προδιαγραφές για τα, για τα τρόφιμα. Βεβαίω πρέπει να αγοράζουμε από τη Δανία, τη Γερμανία και άλλες ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν ακολουθούν τα ίδια κριτήρια ε, στα οποία έχουμε συμφωνήσει και τους ίδιους όρους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να διακρινίσουμε αυτό το σημείο ε, και σε επίπεδο εθνικών διαλόγων, γιατί σε πολλές φορές στους δημόσιους διαγωνισμούς, ε, στους για δημόσιες προμήθειες για τα τρόφιμα, ε, παίρνουν μια ιδιαίτερα συναισθηματική τροπή. Επίσης συμφωνώ ότι πρέπει να έχουμε αυτό το value for money, όχι μόνο δηλαδή να εστιάζουμε στον οικονομικό παράγοντα, αλλά πρέπει να καθορίσουμε και τι είναι αυτό το, η σχέση ποιότητας και τιμής, να το προσδιορίσουμε. υπάρχουν και τοπικά προϊόντα, τα οποία όμως που δεν λαμβάνουμε τόσο πολύ υπόψη αυτόν τον παράγοντα, γιατί ο τομέας των μεταφορών δεν είναι και το κρισιμότερο ε, πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Εγώ υπέβαλα μια τροπολογία και χαίρομαι που η συγγήτρια ε, την ε, έλαβε υπόψη. Ειδικά από αυτού για τις δημόσιες προμήθειες στον τομέα των τροφίμων, για τα σχολεία, για τα νοσοκομεία και τους οίκους ευγυρία. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι αυτό που είπε ο Σοσιαλδημοκράτης συνάδελφος. Ε, να μειώσουμε την γραφειοκρατία, να απλοποιήσουμε τους κανόνες, να παράσχουμε ευελιξία και ε, να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ποιότητα από πλευρά επιχειρήσεων, όπω κάνουν και οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ισότιμη πρόσβαση στην αγορά. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε διαφορετικού ε, κανόνε, όπω υπόθηκε προηγουμένω, αλλά ε, ίσε ευκαιρίε για πρόσβαση σε αυτή την αγορά. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Ο κύριος Κρίστερς από την Αυστρία. Ευχαριστώ το θέμα της, των κριτηρίων αξιολόγησης ή του χαμηλότερου μειοδότη είναι τόσο παλιό όσο και η πρώτη συζήτηση σε πολλές χώρες γίνεται τώρα ένας διαχωρισμός μεταξύ του χαμηλότερου και του, της υψηλότερης προσφοράς και πολλές φορές η επιλογή δεν δίνεται σε οικονομικά κριτήρια τόσο όσο σε κοινωνικά, περιβαλλοντικά κλπ. Γι' αυτό συμφωνώ πολύ και με αυτά που είπε ο κύριος Κρότσμα. Πρέπει να έχουμε ποιοτικά κριτήρια ε, που πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτά τα, την κοινωνική πτυχή για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε μια σωστή αξιολόγηση των μη οικονομικών κριτηρίων. Πώς γίνεται η επιλογή ε, εκτός οικονομικών κριτηρίων για να εμποδίσουμε και όλες τις προσφυγές που ενδέχεται να γίνουν μετά από την ανάθεση. Άρα λοιπόν ελαστικότητα, απλούστευση ε, εδώ υπάρχει και ένα αμφιλεγόμενο θέμα με την ε, νομική ασφάλεια. Αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς στο νομικό πλαίσιο, υπάρχει νομική ασφάλεια, πρέπει να φροντίσουμε την ελαχιστοποίηση των ε, προσφυγών για παραβίαση των διατάξεων, διαφθορά κλπ. Πολλές φορές, αν εφαρμόζουμε μία ελαστικότητα στις διατάξεις, ε, δημιουργούμε δυσκολίες στην απλώστευση, στην απλοποίηση, ιδίως στο θέμα της κλήρωσης. Ε, αν αυξήσουμε τη χρήση των κληρώσεων, οι υπηρεσίες οι οποίες προκυρήσουν το διαγωνισμό βρίσκονται πολλές φορές σε δύσκολη θέση να εξηγήσουν πώς κατέληξαν και ποιοι συμμετέχουν στην κλήρωση. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρη η διαδικασία της κλήρωσης. Ε, όσον αφορά τώρα τις μικρομεσαίες, πολλές φορές έχουν μία μυρολατρεία και πιστεύουν ότι είναι τόσο δύσκολη και δαπανηρή διαδικασία συμμετοχής που, που δεν αξίζει τον κόπο να συμμετάσχουν. Πρέπει λοιπόν να καθησυχάσουμε τους φόβους τους και να τους δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής. Ε, στην Αυστρία από το 2001 υπάρχει μια υπηρεσία δημοσίων διαγωνισμών για όλη τη χώρα, η οποία συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες ανάγκης δημοσίων προμηθειών και συνεχεία προκυρήσει του διαγωνισμούς. Και είναι μια υπηρεσία η οποία λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια και προσέχει πάρα πολύ και το οικονομικό σκέλος πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία δημοσίων διαγωνισμών δεν θα πρέπει να είναι εχθρική, δεν θα πρέπει να την πολεμήσουμε, αλλά η η υπηρεσία μας αυτή στην Αυστρία, εκτός από την προκήρυξη και ανάθεση, δημιουργεί και διάφορες ημερίδες πληροφόρησης, ενημέρωσης των πολιτών, όπου όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες συμμετοχής. Ε, το θέμα είναι, για τους μικρομεσαίους πρέπει να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν τη φοβία που έχουν, ε, αυτό το βάρος που αισθάνονται, το πλάκωμα αν θέλετε δηλαδή, ότι είναι τρομερό, τρομερά δύσκολη συμμετοχή σου σε δημόσιους διαγωνισμούς. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής, Σανγκάλη από την Ιταλική Γερουσία. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για όλη αυτή την εργασία. Τάχιστα θα ασχοληθώ με το θέμα της μικρομεσαίας επιχείρησης, όπως άλλωστε έκαναν και αρκετοί συνάδελφοι θα προσπαθήσω να χαράξω συγκεκριμένους προσανατολισμούς προς την κατεύθυνση αυτή. Δυσκολεύονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην Ιταλία αλλά και αλλού στις ε, δημόσιους διαγωνισμούς ε, και οικονομικού χαρακτήρα βέβαια. Θα πρέπει όπως το είπαμε να υιοθετήσουμε εργαλεία και οικονομικές μεθόδους ε, για να μπορούν να χρησιμοποιηθεί ακριβώς κεφάλαιο κινδύνου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτούς διαγωνισμούς με μια εγγύηση και από πλευράς κράτους για αυτές τις επιχειρήσεις και επίσης η αποπληρωμή απέναντι στους ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στη χώρα μου καθυστερούν ιδιαίτερα τις πληρωμές τις καθυστερεί το δημόσιο γι' αυτό χρειάζεται μια άσκηση πίεσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για, τις, για γρηγορότερες πλήρωνες και επίσης ε, από την άλλη μεριά ε, μεγάλες επιχειρήσεις ε, ευνοούν, αλλά θα πρέπει να ευνοηθούν οι μικρές να μεγαλώσουν και επίσης όπως στις ΗΠΑ Πολιτείες της Αμερικής θα πρέπει να υπάρχει μια ποσόστοση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε διάφορου τομείς και σε διάφορους, ε, διάφορα έργα ανεξάρτητα από το ΑΕΠ τους. Και επίσης χρειάζεται μια ρύθμιση για την πρόσβαση στους διαγωνισμούς αλλά για ένα πραγματικό ανταγωνισμό θα πρέπει να δούμε τους τρόπους επιλογής των επιχειρήσεων και σε σχέση με τα όσα στοιχείουν ε, και θα πρέπει να αποφύγουμε την ανάμειξη εγκληματικών οργανώσεων είτε μη εντελώς διάφανων επιχειρήσεων και επίσης βλέπουμε ότι στις κατασκευές κερδίζουν εταιρείες αυτούς τους διαγωνισμούς που δεν είναι οικοδομικές εταιρείες αλλά είναι οικονομικές και μετά τα δίνουν υπεργολαβία. Η υπεργολαβία θα πρέπει κατάλληλα και ακριβώς να ελέγχεται. Και επίσης η παρέμβαση υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο διαδίκτυο που με κάποιες οικονομικές ευκολύσεις να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε υψηλότερου ποσού διαγωνισμούς θα ήταν κάτι το θετικό και έτσι να μπορούν αυτές οι επιχειρήσεις να συμμετέχουν όπως πρέπει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και η κυρία Γκέπχαρτ, καταρχά. Τελευταίοι δύο μιλητέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Σενγκάλη, θα κάνω μια προκαταρτική παρατήρηση. Πριν, ε, πρόσφατα ε, υιοθετήσαμε ένα νομοθέτημα το οποίο πρέπει να μεταφερθεί ακόμα στα εθνικά δίκαια, το οποίο κάνει ακριβώς αυτό το οποίο εσείς ζητάτε. Είναι καθοδόν δηλαδή Η κυρία Βάιλερ ήταν η συγγήτρια αυτής της έκθεσης νομοθετικού περιεχομένου. Αν θέλετε πληροφορίες απευθυνθείτε σε εκείνη. Εγώ όμως είχα ζητήσει το λόγο αυθόρμητα για ένα άλλο θέμα. Δεν είχα πρόθεση να μιλήσω, αλλά ήθελα να πω κάτι μεταξύ των προσφορών της χαμηλότερης τιμής και της βέλτιστης αξίας από το 2004 είχαμε ζητήσει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη η καλύτερη προσφορά έναντι της φθηνότερης. Διότι πάντοτε λέγαμε πρέπει πάντοτε να χειριζόμαστε λογικά και σωστά τα χρήματα των φορολογούμενων. Άρα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την ποιότητα και όχι μόνο τη φτύνια. Διότι το, ένα έργο, ένα πρόγραμμα ας πούμε είναι μακροπρόθεσμο ε, γίνεται για πολλά χρόνια. Επίσης πρέπει να φροντίσουμε τη σωστή πληρωμή ε, των εργαζόμενων, τη σωστή αμοιβή. Και πολλές ε, φορές βλέπουμε ότι στα φτηνότερα έργα, στις φτηνότερους διαγωνισμούς και οι αμοιβέ ε, πέφτουν κάτω από το παραδεκτό κοινωνικό επίπεδο. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα κοινωνικά κριτήρια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τη βέλτιστη προσφορά, για τη βέλτιστη προσφορά και να σκεφτόμαστε μεσοπρόθεσμα και βράχη πρόθεσμα και, όχι, και μακροπρόθεσμα, συγγνώμη, και όχι μόνο με βραχή πρόθεσμη προοπτική αύριο μεθαύριο. Λοιπόν, ε, γι' αυτό όταν επιτύχουμε να εφαρμόσουμε μία μέθοδο που θα επιλέγει την καλύτερη προσφορά θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο στόχο μας μακροπρόθεσμα έργα και έργα ποιότητας. Μην ξεχνάμε τη μελλοντική εικόνα. Δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε μέσω άλλων υπεργολάβων να υπονομεύεται μια σωστή επιλογή και να εφαρμόζονται τελικά αρνητικά κριτήρια. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Uh, Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Όλα αυτά τα θέματα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και βεβαίως έχουμε κάνει και πολλή δουλειά πάνω σε αυτό στην Επιτροπή μας. Η κυρία Ροζοτιούν έχει τον τελευταίο λόγο. Ευχαριστώ. Όχι, μετά. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ την κυρία Ρούλε για αυτή την έκθεση. Θα μιλήσω πολωνικά. Η, κυρία Ρούλε, όπως και πολλοί άλλοι ομιλητές ε, σήμερα και χτες, αναφέρει φέρθηκαν στο φόρουμ αυτό στην Κρακοβία που μας ενέπνευσε για τη σημερινή μας δουλειά. E, και πιστεύω ότι θα πρέπει τώρα να φροντίσουμε να συνεχίσουμε αυτές τις ε, συζητήσεις, τις κοινέ συνεδριάσεις μαζί και με εμπειρογνώμονες του τομέα. Εγώ δεν ε, έλαβα μέρος στην μερίδα εργασίας ε, που ανέφερε η Χάιντι Ρούλε γιατί έμεινα εκεί που συζητούσαν τις ε, δημόσιες, ε, τους δημόσιους διαγωνισμούς. Όμως ήθελα να σχολιάσω λίγο αυτά, αυτά τα κριτήρια του, του φθηνότερου ε, μειοδότη ή του καλύτερου. Όταν μιλάμε για δημόσιους διαγωνισμούς όλοι έχουμε κάποια προσωπική εμπειρία. Όπως ξέρετε η Πολωνία αυτή τη στιγμή κατασκευάζει πάρα πολλούς δρόμους, πάρα πολλές ε, οδικά δίκτυα και τα κριτήρια όλα αυτά και οι δημόσιοι διαγωνισμοί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τους επενδυτές διότι υπάρχει μεγάλο κόστος ε, στην ποιότητα ε, και, και, και, και όλοι ενδιαφέρονται πολύ έντονα για αυτό το θέμα που συζητάμε εδώ. Αναφέρεται, επίσης αναφέρεται καθόλου το, το θέμα των έκτακτων παροχών. Μιλάμε συνέχεια για διαφάνεια, αλλά οι έκτακτες ε, παροχές, ε, τα concessions δεν αποτελούν μέρος των δημοσίων διαγωνισμών και γι' αυτό η Κομισιόν πρέπει να ε, δημιουργήσει, να, να κάνει ορισμένες προτάσεις και γι' αυτό το θέμα. Έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή προτάσεων της Κομισιόν. Και πολλές ε, τοπικές κοινότητες ε, ε, υποφέρουν διότι δεν τους αναθέτονται δημόσια έργα λόγω των εξαιρέσεων που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Ανάθεσης. Μην ξεχνάτε ότι οι εξαιρέσεις μπορούν να αυξήσουν και τον ανταγωνισμό και δεν είναι ένα τόσο κακό στοιχείο όπως πολλοί θεωρούν. Ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι ιδιαίτερα που είχατε τον τελικό λόγο διότι είσαστε ενεργό μέλος της Επιτροπής μας. Τρία λεπτά τώρα στην εισηγήτρια για να ολοκληρώσει. Και να μας πει ποιο θα είναι το επόμενο βήμα της έκθεσης και πώς θα ενσωματωθεί στην ομοθεσία. Ε, να μας πει και για το χρονοδιάγραμμα, για το μέλλον δηλαδή της ε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Ευχαριστώ όλους όσους ε, σχολίασαν και όσους μίλησαν. Τον Οκτώβριο θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια η έκθεσή μου. Μετά περιμένουμε τις προτάσεις της Κομισιόν το Δεκέμβριο. Η Κομισιόν μας είπε ότι θα μας παρουσιάσει ένα πακέτο για την νέα επεξεργασία όλου του πακέτου θα έχει τρία τμήματα. Καταρχάς αναθεώρηση της οδηγίας ανάθεσης, δεύτερον προσφορά υπηρεσιών και τρίτον αμοιβαιότητα. Ε, δηλαδή ε, πώς θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα των αθέμητων προσφορών και διαγωνισμών. Αυτά, αυτά ως προς το πακέτο της Κομισιόν. Τώρα, όσον αφορά Αυτές τις εξαιρέσεις ε, πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο είχε μία ιδιαίτερη ε, θέση και πιστεύει ότι αυτές οι ε, κατεξαίρεση παραχωρήσεις είναι ένα αρνητικό στοιχείο διότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι που εφαρμόζονται αυτές οι κατεξαίρεση παραχωρήσεις δεν μπόρεσε η Κομισιό να μας αποδείξει ότι ακριβώς ποιες τρευλώσεις εννοεί η Κομισιόν ε, σε αυτές τις έκτακτες παραχωρήσεις. Η Κομισιόν μας είπε ότι μέσα στην αναθεώρηση θα εξηγήσει περισσότερο το καθεστώς αυτό των concessions, των παραχωρήσεων. Ε, ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το ίδιο πράγμα αυτές οι έκτακτες παραχωρήσεις με τους δημόσιους διαγωνισμούς. Μας έχουν εκπαιδεύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι και ένα στοιχείο που δυσκολεύει τη σωστή συνεργασία και την ομαλή διαχείριση των διαγωνισμών. Τώρα, ποια είναι, σαφώς υπάρχει σχέση μεταξύ δημοσίων προκηρύξεων και ανατομίας και αηφόρου ανάπτυξης. Βεβαίως υπησέρχεται και το στοιχείο της επικουρικότητας ε, στα κράτη-μέλη. Οι Σουηδοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο θέμα της προστασίας της ευζοίας των ζώων. Η ευζοία των ζώων εξαρτάται περισσότερο από τον τρόπο παρασκευής, ας πούμε, ενός προϊόντος, του κρέατος και όχι στο προϊόν αυτό αυτό. Πρέπει όμως και στις παραγωγικές μεθόδους ε, να βρούμε έναν τρόπο να καλυφθούν στις προκηρύξεις προμηθειών από τα πρώτα βήματα, δηλαδή στις τεχνικές προδιαγραφές προκήρυξης ενός διαγωνισμού ας πούμε για προμήθεια κρέατος πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια ευζοίας των ζώων. Ακριβώς αυτό θέλουμε. Όχι μόνο να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο προϊόν, αλλά και στις προηγούμενες και προκαταρτικές φάσεις ε, ε, παραγωγής. Ε, συμφωνώ απόλυτα ε, με αυτά που είπε ο Αυστριακός συνάδελφος για την απλούστευση, απλοποίηση των διαδικασιών και περισσότερη ενημέρωση και πληροφόρηση. λιγότερο χαρτοβασίλειο, λιγότερα έγγραφα και τεκμηρίωση που χρειάζεται, όλα αυτά να τα απλουστεύσουμε. Και τέλος, διαφθορά. Η διαφθορά και εδώ ακούσαμε, σημαντικές, ε, έγιναν σημαντικές παρατηρήσεις το πώς η διαφθορά υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα και τη διαφάνεια, το θέμα των υπεργολάβων και υπεργολαβιών. Δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες ακόμα μεταξύ των κρατών μελών στο θέμα της διαφοράς, διαφθοράς. Συγγνώμη. Και αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε. Καλύτερη ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών. Σας ευχαριστώ, κυρία που Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ε, να μας κρατήσετε ενημερούς στη συνέχεια. Περνάμε τώρα στο τελευταίο τμήμα της συνεδρίασής μας. Εδώ εμείς οι τρεις πρόεδροι είμαστε το μοναδικό εμπόδιο που έχετε ε, για το μεσημεριανό γεύμα. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ξεκινώντας θα δώσω το λόγο στους ε, συμπροέδρους ε, από την ε, Πολωνική Γερουσία. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι ήταν με ιδιαίτερη χαρά εργάστηκα και με τους δύο και θεωρώ ότι η συνεργασία μας με την Πολωνική Προεδρία στο σύνολό τη ήταν πολύ θετική. Σε σημεία, ε, στα θέματα της ε, ενιαίας αγοράς, η Προεδρία έδειξε πραγματικό ενδιαφέρον και αυτό ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για μας και για σας ελπίζω ως μέλη του Εθνικού Κοινοβουλίου που ε, ήρθαν εδώ. Και είναι πολύ σημαντικό ε, που διοργανώθηκε αυτό το Single Market Forum στην Κρακοβία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και πράγματι αποτέλεσε ευκαιρία για να διεξαγάγουμε μια πολύ ε, χρήσιμη και επικοδομητική συζήτηση μαζί σας. Πέρα από αυτό, υπήρξε ε, και μια εκδήλωση στην κεντρική πλατεία της Χαρκοβίας ε, και οι πολίτες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια Κυριακή απόγευμα, ήρθαν εκεί για να μάθουν τι ακριβώς μπορεί να προσφέρει σε αυτούς η ενιαία αγορά. Και μία από τις αποστολές μας ε, σε αυτή την επιτροπή ήταν η ενιαία αγορά να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των καταναλωτών. Αυτό ήταν και ο στόχο πίσω από το Single Market Act ε, και προσπαθεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες και τα συμφέροντα των καταναλωτών. για να γίνει αυτό θα πρέπει σίγουρα να αναλάβουν δράση και τα εθνικά κοινοβούλια, να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίω όλοι πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλέ ε, ευκαιρίε που δεν έχουμε αξιοποιήσει ακόμα, ευκαιρίε για τους πολίτες να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην ενιαία αγορά, αλλά και να αποκομίσουν κέρδη από αυτό αλλά και για τους πολίτες, τα ωφέλη που έχουν ε, στις ε, διασυνοριακές τραπεζικές αλλαγές και ο ρόλος μας είναι να τους ε, παράσχουμε ξεκάθαρες πληροφορίες και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το διαδίκτυο και την πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες αυτός ο στόχος θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της ενιαίας αγοράς. Ε, Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των πολιτών είναι ότι τους δίνουμε πρόσβαση να, ε, να, να, βρουν όλα αυτά τα εμπορεύματα και, και τα λοιπά, αλλά υπάρχουν άλλα προβλήματα μετά που δεν τους αφήνουν ουσιαστικά να τα απολαύσουν. Παρομοίως, Πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε τα μέσα για τα εργαλεία της ενιαίας αγοράς, ε, οι δημόσιες προμήθειες και η ε, αμοιβαία αναγνώριση επιστοποίησης είναι δύο από τα κύρια εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ενιαία αγορά. Ανακούσαμε αν ακούσαμε τις απόψεις σας, μας είπατε τους προβληματισμούς σας. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε δράση Και μία από τις πρωτοβουλίες αυτής της Επιτροπής είναι να κάνει το ε, πολιτικό έργο πριν λάβουμε νομοθετικό, νομοθετική πράξη από την Επιτροπή. Θέλουμε δηλαδή να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος, όχι μόνο να υποβάλουμε τροπολογίες. Γι' αυτό και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει περισσότερα και χαίρομαι που ε, οι συνάδελφοί μου και οι συντονιστέ όλων των ομάδων ήταν εδώ σήμερα και χαίρομαι γι' αυτό. Συμφώνησαν να συνεργαστούμε και βλέπουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν με θετικό βλέμμα αυτή την ε, πρωτοβουλία. Γι' αυτό και εμείς έχουμε πολλές ε, επαφές και συνεδριάσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Όπως είπα και προηγουμένως, εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας και στις ε, επιτροπές να, να έρθουμε εδώ ακόμα και να, να συνεδριάζουμε μέσω τηλεδιασκέψεων και όλα αυτά. Θέλουμε να μιλήσουμε με τις επιμέρους χώρες και με τρίτες χώρες για την ενιαία αγορά. Θα πάμε στην Τουρκία σύντομα, θα μιλήσουμε με τους Τούρκους συναδέλφους και στην Κροατία θα πάμε και στη Δανία ε, ως επερχόμενη Προεδρία ε, με στόχο να συνεχιστεί το έργο της Πολωνικής Προεδρίας. Ελπίζω λοιπόν, σας ευχαριστώ αρχικά για την ενεργό συμμετοχή σας και τις εξαιρετικές σας παρεμβάσεις και που συμμετείχατε με σοβαρότητα σε αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω λοιπόν να μεταφέρετε και να μεταβιβάσετε αυτό το μήνυμα στα εθνικά σας κοινοβούλια. Ήταν τιμή μου ε, που συμπροέδρευσα αυτής της ε, συνεδρίασης. Ελπίζω στην επόμενη συνεδρία να βρισκόμαστε σε αίθουσα που να παρέχει και τσά και καφέ και καλύτερε υπηρεσίε. Ωστόσο, είχατε την ευκαιρία να πάρετε το λόγο εδώ. Ε, ίσως η απευθεία σύνδεση να μην ήταν τόσο καλή όσο άλλες φορές, γιατί δείχνει ε, μια ευρύτερη εικόνα και όχι τους μεμονωμένους ομιλητές. Ελπίζω σύντομα να λάβετε και την ε, έκθεση, αυτή την ομοδότηση μάλλον. Και όπως ε, είπα, παρακαλώ, συνεχίστε να ε, είστε σε επικοινωνία και σε επαφή μαζί μας, ούτω ώστε να γίνετε φίλοι, να, μάλλον να, να ζητήστε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο τη ΕΜΚΟ για να έχετε έτσι όλες αυτές τις πληροφορίες σχετικά με τι εργασίε μα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν που ήρθατε εδώ σήμερα και εν κατακλείδη θα ήθελα να πω ότι μας ευχαριστεί ιδιαίτερα που ε, η Γερουσία και η ΣΕΜ επέλεξαν την, το θέμα της ενιαίας αγοράς ως ε, κύριο θέμα. Χαίρομαι που αναλάβατε αυτή την πρωτοβουλία λοιπόν. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μπρεβίνσκι και Τρίνσκι για τις, ε, κατα... τις τελικές τους παρατηρήσεις. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, θερμά. Όπως μόλις αναφέρατε, Έχουμε ακόμα, πρέπει όλοι να υπομείνουμε ακόμα δύο παρεμβάσεις πριν από το γεύμα. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να εκφράσω είναι η μεγάλη μου ικανοποίηση για αυτή τη συζήτηση. Άκουσα πάρα πολλές ε, λεπτομέρειες, πολλά στοιχεία για το τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον και όταν γυρίσουμε πίσω στην Πολωνία, τι θα πούμε στους πολίτες μας εάν τους πούμε όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε και όλα αυτά τα προβλήματα που εντοπίσαμε και πρέπει να λυθούν, πιστεύω ότι θα έχουν την, την, την αίσθηση ότι η κατάσταση είναι χαόδης. Για να αποφύγουμε λοιπόν αυτή την εικόνα, θα σας εξηγήσω τι θα πω στην Πολωνία όταν γυρίσω. Μελετώντας τις ρίζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαβαίνω ότι πρέπει να επιλέξουμε τη μελλοντική μας πορεία. Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Ή θα επικεντρωθούμε μόνο στις εθνικές προτεραιότητες ή θα δείξουμε το θάρρος που χρειάζεται για να συνεργαστούμε για ένα κοινό μέλλον έχτες άκουσα από εσά ότι σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν έντονες ανησυχίες για το μέλλον της ενιαίας αγοράς, της κοινή αγοράς. Ανησυχίες επίσης για την αγορά εργασίας και τις ε, στρεβλώσεις της. Βλέπω λοιπόν σαφώς ότι υπάρχει βούληση για θετική δράση και για την ε, εφαρμογή αλλαγών για να γίνουν πολλές αναγκαίες αλλαγές. Διάβασα μια φορά ότι εάν θέλεις να επιβιώσεις αν θέλεις να μεταναστεύσεις σε, μια άγνωστη χώρα, μην ε, χτίσεις πρώτα ένα πλοίο για να πας, αλλά πήγαινε πρώτα στην άγνωστη αυτή χώρα για να δεις πώς είναι και, και τι χρειάζεται. Ε, εμείς ξέρουμε λοιπόν τι χρειάζεται για το μέλλον είναι άγνωστο το μέλλον, αλλά ξέρουμε τι χρειάζεται. Καλύτερη διαχείριση, καλύτερη δίκηση, μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη σαφήνεια. Και κάτι άλλο που ανέφεραν οι Σκανδιναβοί φίλοι. Πολλές φορές όταν φυσάει ένας δυνατός άνεμος, ορισμένοι χτίζουν ένα τείχο προστασίας. Άλλοι όμως χτίζουν ανεμόμυλους για να τους χρησιμοποιήσουν για ενέργεια. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάθε στοιχείο μπορεί να ερμηνευθεί και θετικά και αρνητικά. Εδώ προερχόμαστε όλοι από διαφορετικά παρελθόντα, από διαφορετικούς, ε, διαφορετικά πολιτιστικά ας πούμε, ε, παιδεία, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλοι μας την εμπειρία για το κοινό όφελος. Ε, μην ξεχνάμε και το, την καινοτομία, της ε, της νέες ανακαλύψεις, τη νέα τεχνολογία. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μου δώσατε την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτήν την ε, ηλεκτρονική συζήτηση και Ευχαριστώ και τον Πρόεδρο που μας ευχαρίστησε, αλλά και εγώ τον ευχαριστώ θερμά για τη διεξαγωγή αυτής ε, της ε, συνεδρίασης. Έκανε μια θαυμάσια προπαρασκευαστική εργασία. Ήρθαμε λοιπόν εδώ πολύ καλά προετοιμασμένοι και όλη η διαδικασία των δύο ημερών εξελίχθηκε πάρα πολύ ομαλά και εύχομαι σε όλους καλή επιστροφή στις πατρίδες τους και καλή αντάμωση. Ε, Ευχαριστώ και εγώ κυρίες και κύριοι. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα μιλήσω και ο πιο σύντομος. Ο, κύριος, ο πρόεδρος Χάρμπορ ε, ε, παρουσίασε πάρα πολύ καλά τα συμπεράσματα αυτής της κοινή συνεδρίαση. αυξήσαμε τον κύκλο των φίλων μας ε, από την ΙΜΚΟ και μας εντυπωσίασαν ιδιαίτερα οι παρεμβάσεις και οι εργασίες. Όπως είπε και ο συνάδελφός μου ο κ. Ε, Ταβίνσκι, ε, ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την πρωτοβουλία αυτή που της Πολωνικής Προεδρίας και του Προέδρου Χάρμπορ μια κοινή πρωτοβουλία Προεδρίας και Επιτροπή ΣΥΜΚΟ για τη διεξαγωγή αυτής της, αυτών των συνεδριάσεων. Ε, μέσα σε μία εβδομάδα λάβαμε μέρος σε δύο πολύ σημαντικές ευρωπαϊκές συνεδριάσεις με δύο πολύ επίκαιρα θέματα. Ε, η πρώτη συνεδρία έγινε στην Κρακοβία, μία από τις παλιότερες ευρωπαϊκές πόλεις και η δεύτερη συνάντηση εδώ στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, όλοι μας ε, και μιλώ εκ μέρους όλων των μελών της πολωνικής αντιπροσωπείας ως όλοι που, εμείς που θα επιστρέψουμε στα εθνικά μας κοινοβούλια και όσοι επανεξελέγησαν για την επόμενη σητεία μετά τις εκλογές της Κυριακής σκληρά στις επιτροπές τους και ειδικά στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ε, για την ανάπτυξη και βελτίωση της ε, ενιαίας αγοράς η ευρωπαϊκή αλλά και η εθνική διάσταση θα την έχουμε πάντα κατά νου, θα την έχουμε πάντοτε υπόψη και θα επωφεληθούμε των δικών σας προτάσεων και ιδεών για τη δική μας εργασία στην Πολωνία. Ε, έχουμε εξαιρετική Ακούς ε, πρέσβεις, την κυρία Χάντλικ, την κυρία Ρουρατούν, τον κύριο Τσασκόφσκι. Έχουμε εξαιρετικούς Πολωνούς ε, βουλευτές συγγνώμη, και εκπροσώπους εδώ, τους οποίους ακούσαμε και τους εκτιμούμε ιδιαίτερα στην Πολωνία και είναι και οι εκπρόσωποι μας, οι πρέσβεις μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ενιαία αγορά είναι ένα τεράστιο ευρωπαϊκό έργο ένα τεράστιο τομέα τον, τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας γιατί θα είναι καθοριστικός για το μέλλον μας. Συμπεραίνοντας και ολοκληρώνοντας θέλω να εκφράσω μία ευχή ότι αυτό το πρόγραμμα μετά από όλες αυτές τις προσπάσεις που κάνουν τα τρία θεσμικά όργανα και τις δικές σας προσπάσεις κύριε Πρόεδρε Εύχομαι το, το έργο αυτό το μεγάλο να επιτύχει και να ωφελήσει όλους τους πολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει λοιπόν, Επομένως κλείνουμε εδώ τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή διαμονή στις Βρυξέλλες, να μείνετε εδώ και καλή επιστροφή. Hello. Thank you very much.